Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους ε, σε αυτή την ε, κοινή συνεδρίαση δύο επιτροπών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Επιτροπής ΕΚΟΝ και της Επιτροπής ΡΕΤΖΙ. Οργανώνεται η συνεδρίασή μας λόγω της ακρόασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναστολή τον ε, ΔΕΗ, μέρο του διαθρωμένου διαλόγου που προβλέπει το άρθρο 23, παραγωγός 15 του Κοινωνισμού 1303-2013. Καταρχήν, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Γεωργία Κατάνοη και την Επιτρόπο Κορίνα Κρέτσου στη σημερινή μα συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε για την έλευσή σας εδώ και για τη μελλοντική σας συμμετοχή. Για πρώτη φορά Συνεδριάζουμε σήμερα σε αυτό το μορφότυπο για να ξεκινήσουμε τον πρώτο διαρθρωμένο διάλογο με την ακρόαση με την Κομισιόν για την πιθανή αναστολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Ξεκίνησε η διαδικασία αυτή τον Ιούλιο όταν ε, το Συμβούλιο ε, είδε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν είχαν αναλάβει αποτελεσματική δράση για να μειώσουν τα ελλείμματά τους ε, κάτω από την τιμή αναφορά ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής σε δυνάμει ε, του Συμφωνού Σταθερότητας και ανάπτυξη, ε, Έτσι λοιπόν η απόφαση του Συμβουλίου πρόβλεψε κυρώσεις υπό τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. Τα κυρία στοιχεία ήταν ε, μια πιθανή επιβολή προστήμων και η αναστολή των πληρωμών ή των πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων δυνάμει των διαφορετικών και επενδυτικών ταμείων σε αυτά τα δύο κράτη-μέλη. Τον Αύγουστο αποφασίστηκε το Συμβούλιο ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα στι δύο χώρε. Η Κομισιόν τώρα πρέπει να παρουσιάσει στο Συμβούλιο μία πρόταση να αναστείλει ένα μέρο ή όλε τι πληρωμέ ή τι πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων για τι δύο χώρε σε σχέση με τα διαφορετικά ταμεία. Όμως, ε, υπό την σημερινή νομοθεσία, η Κομισιόν μπορεί να κάνει μια τέτοια πρόταση μόνο μετά από διαρθρωμένο διάλογο με το Κοινοβούλιο. Επομένω, σήμερα έχουμε συναντηθεί εδώ για να ξεκινήσουμε αυτό το διάλογο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι απόψε μαζί μας ε, είναι και εκπρόσωπος της Επιτροπής των Περιφερειών ε, που έχει δημιουργήσει ε, ουσιαστικά ε, μια ειδική θέση για την κατάσταση στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Μπορείτε να δείτε και την ιστοσελίδα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη για τα εισαγωγικά του σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο Κατάνων και την Επίτροπο ε, Κρέτσου για αυτό τον διευθυντικό διάλογο. Νομίζω ότι πολύ σωστά συνοψίσατε ε, το διαδικαστικό και νομικό βήμα που μας οδήγησε να εκινήσουμε αυτό τον ιδιωτικό διάλογο. Επομένω, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι με αυτή την ε, συνεδρίαση ξεκινούμε λοιπόν αυτόν τον διαδικαστικό διάλογο και θα εξετάσουμε κατά πόσο θα κάνουμε και περαιτέρω βήματα και ποια θα είναι αυτά βάσει και των αποτελεσμάτων ε, του διαδικαστικού διαλόγου που όπως ξέρετε θα αξιολογηθεί στη συνέχεια από τι συνδυάσεις των συντονιστών των δύο επιτροπών. Επομένω, δεν μπορούμε ακόμα να γνωρίζουμε κατά πόσο θα ολοκληρώσουμε αυτή τη δικασία σήμερα ή όχι. Ένα δεύτερο σχόλιο το οποίο θεωρώ σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα σαφές στοιχείο του νομοθέτη ότι θα υπάρξει επανεξέταση που προβλέπεται βάσει του κανονισμού για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Όμω, όπω είπε και συνάδελφο, υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη δύο διαφορετικών διαδικασιών που και οι δύο κινούνται βάσει απόφαση του Συμβουλίου. Ε, αποφασίζει λοιπόν το Συμβούλιο ότι δεν έχει υπάρξει διορθωτική ενέργεια, όμω κατόπιν ε, πρόταση τη Επιτροπή, το Συμβούλιο αποφάσισε να ακυρώσει τα πρόστιμα προ τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντα υπόψη ε, τι εξαιρετικέ οικονομικέ ε, συνθήκε, αλλά και τι τις δεσμεύσεις, αλλά και τις ενέργειες που λαμβάνουν τα δύο κράτη-μέλη. Από την άλλη, έχουμε αυτό το δεύτερο στοιχείο, που καλύπτεται από τον ε, κανονισμό που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση. Βέβαια, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει πλήρω υπόψη τα αποτελέσματα του τεχνικού διαλόγου, τη απόψη του Κοινοβουλίου δηλαδή, αλλά και ένα άλλο μακροοικονομικό στοιχείο. Θα έχουμε λοιπόν ε, χρόνο να τα συζητήσουμε επί τη ουσία. Ποιο είναι δηλαδή ε, το η διακριτική ευχέρεια ε, που ίσως να είναι μεγαλύτερο από αυτό που θεωρεί η Επιτροπή. Ακριβώς αυτό θα συζητήσουμε εδώ. Υπενθυμίζω τέλος ότι μία από τις αιτίε αυτού του διαλόγου είναι ακριβώς για να έχουμε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση τεκμηριωμένη για τα βήματα που θα ληφθούν. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτέ τι λεπτομερεί αναφορέ. Αν δεν τι ακούσουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τον διευθυντικό διάλογο. Παρακαλώ, έχετε και πάλι το λόγο. Ο, η πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, να δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από ό,τι ξέρω, βάσει προγράμματος. Ο κύριος Κατάινεν έχει πρώτο το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε και κύριε Κουαλτήρη, που μας καλέσατε στην ακρόση αυτή ή στην ανταλλαγή απόψε. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ σήμερα για να ακούσουμε τις απόψεις σας και να δώσουμε διευκρινήσεις ε, σε σχέση με τη λειτουργία τη μακροοικονομική αρεσιμότητα των διαθερωτικών και επενδυτικών ταμείων. Αυτό δεν έχει να κάνει ιδιαίτερα με το σύμφωνο σταθερότητα. Υπάρχει ένα σύνδεσμο, αλλά περισσότερο είναι θέμα μακροοικονομική αρεσιμότητα των ταμείων ΕΣΥ, όπως ξέρετε, δεσμεύεται η Κομισιόν ε, να ε, παρά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει και επενδύσει για να έχουμε ανάπτυξη και θέσει εργασίας. Επίση δεσμευόμαστε στην κοινωνική δικαιοσύνη και είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε φιό του κανόνες για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ο λόγος που είμαστε εδώ απόψε οφείλεται στην υιοθέτηση από το Συμβούλιο στις 12 Ιουλίου φέτος δύο αποφάσεων που μιλούσαν για την ε, αναποτελεσματική δράση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, για τα έτη 2013-2015. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν αναγνωρίζει ε, το ότι πρέπει να ε, δούμε ε, ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν ε, οδηγηθεί σε δύσκολες διαδικασίες το Συμβούλιο αποφάσισε στις 8 Αυγούστου να μην επιβάλλει πρόστιμα υπό το διορθωτικό σκέλος του Συμφωνού σταθερότητα και Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα έχουμε έναν διοσυνομικό δρόμο για κάθε χώρα και ζήτησε να υποβάλουν αναφορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για τις δράσεις που έχουν αναλυφθεί. Οι εκθέσεις αυτές ταυτόχρονα ε, θα παρουσιαστούν ως το ε, δημοσιονομικό σχέδιο προπολογισμού. Η ίδια η απόφαση του Ιουλίου ε, δημιουργεί την απόφαση της μικροοικονομικής αιρεσιμότητας που συνδέει τα ε, ταμεία ΕΣΥ και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση όπως έχει συμφωνηθεί από τους συνομοθέτες. Υπό αυτούς τους κανόνες η Κομισιόν πρέπει να προτείνει μια αναστολή ενός μέρους ε, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα ταμεία, των ταμείων για το 2017. Όχι πληρωμές, αλλά πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων μετά από διαρθρωμένο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε πολλές πληρωμές και πόρους διαθέσιμους για τις χώρες αυτές, ακόμη και αν η Κομισιόν αποφασίσει να αναστείλει μέρος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Εγώ έγραψα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις 4 Ιουλίου για να τον ενημερώσω για τη διαδικασία και να εκφράσω την ετοιμότητα της Κομισιόν να συμμετέχει σε ένα διαρθρωμένο διάλογο για την εφαρμογή του μέτρου. Είμαι ικανοποιημένο που μπορούμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων σήμερα, 3 Οκτωβρίου, με τους βουλευτέ διαφόρων επιτροπών. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε του πρόεδρου τη Επιτροπών Ρέτζι και ΕΚΟΝ για τη διοργάνωση της συνεδρίαση αυτής. Αναμένουμε μια ειλικρινή συζήτηση και φυσικά θα αναφέρουμε και το περιεχόμενο της συζήτησης αυτής στους συναδέλφους μας. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Κρέτσου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Και βεβαίως ε, χαιρετίζω και εσά, αλλά και τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική αυτή τη συζήτηση. Είναι και μια ένδειξη του υψηλού σεβασμού που υπάρχει μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Και ε, θα ήθελα να συμπληρώσω τα όσα ανέφερε προηγουμένως ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν και να δώσω περαιτέρω εξηγήσει ε, για τις εξελίξεις αυτές. Όπως έχει δημοθεί βάσει του άρθρου 23 του κανονισμού, όταν ε, το Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι υπάρχει έλλειψη ε, αποτελεσματικής, αποτελεσματικών ενεργειών υπό τα διευθυντικά μέτρα για το ε, Σύμφωνο Σταθερότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει, νομικά δηλαδή είναι δεσμευμένη, να ε, κάνει πρόταση για την μερική τουλάχιστον αναστολή των ε, για την επόμενη χρονιά και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η δυνατότητα να, να ληφθεί αυτή η απόφαση μετά τον ιδρυτικό διάλογο. Είναι ένας πολύ δημοκρατικός τρόπο τρόπος ε, να δράσουμε από κοινού. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι η πιθανή αναστολή ε, των ε, κονδυλίων αυτών των ταμείων δεν είναι κύρωση. Θα ήταν κύρωση υπό το Ταμείο Σταθερότητας που προβλέπει κατευθείαν κυρώσεις. Τώρα πρόκειται για ένα από πολλά μέτρα που συνδέεται με την αιρεσιμότητα, ε, τις ειδικής αναχώρησης συστάσεις και θέτει το σωστό πλαίσιο, ώστε να μεγιστοποιεί το αντίκτυπο των ταμείων. Υπό αυτή την έννοια, ίσως ορισμένοι να ήσασταν και εδώ στο Κοινοβούλιο όταν υιοθετήθηκαν αυτό αυτός ο κανονισμός. Ξέρετε ότι είχε υιοθετηθεί από ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εν είδη νομοθετών. Και θυμάμαι όταν είχε υιοθετήσει στο Κοινοβούλιο την αιρεσιμότητα, είχε ιδωθεί ως μια θετική αιρεσιμότητα, ότι δίνει δηλαδή αρκετό χρόνο ε, στα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις ειδικές αναχώρες συστάσεις εμπροκειμένων. Σας διαβεβαιώ ότι η αναστολή μέρους ε, των διευθυντικών ταμείων δεν έχει καμία βραχυπρόθεσμη επίπτωση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η αναστολή, εάν αποφασιστεί, θα αφορά ένα μερίδιο των χρηματοδοτικών ε, πιστώσεων για την επόμενη χρονιά. Αλλά πίστοση ανάληψης υποχρεώσεων, όχι πληρωμών. Είναι σημαντικό αυτό να το διευκρινίσουμε. Στα διευθυντικά ταμεία έχουμε αυτό τον κανόνα νήσιν 3. Για το 2014, λοιπόν, τα όσα προβλέπονται θα πρέπει να ε, εκταμιευθούν μέχρι το 2017. Εάν, λοιπόν, αναστείλουμε μέρος ε, των πιστώσεων του 2017, θα μας επηρεάσει αυτό μόλις στα τέλη του 2020. Μόνο όμως στην περίπτωση που η εν λόγω χώρα δεν αναλάβει ε, και δεν προβεί σε ενέργειες ε, διορθωτικέ. Σα διαβεβαιώ λοιπόν ότι και οι δύο αυτές χώρες έχουν επαρκείς πιστώσει για τα 14, 15 και 2016 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλει τις πληρωμές για αυτά τα έτη. Γνωρίζουμε ήδη ότι η αναστολή είναι ένα προσωρινό μέτρο. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι το 2020, γιατί ξέρω ότι και οι δύο χώρες έχουν δεσμευθεί να υποβάλουν έως το 15 Οκτωβρίου προσχέδιο προϋπολογισμού. Βεβαίως, η Επιτροπή θα άρει ε, απευθείας ε, τις ε, αναστολές αυτές μόλις συμμορφωθούν οι χώρες αυτές με την απόφαση του Συμβουλίου ή αν το Συμβούλιο θεωρήσει και αποφασιστεί, αποφασίσει ότι έρεται η διαδικασία περιπολικού ελλείμματος. Και μετά θα υπάρξει επαναγραφή στον προπολογισμό αυτών των πιστώσεων και για τις δύο χώρες. Ό,τι αφορά το επίπεδο της αναστολής, τα κριτήρια του κανονισμού ε, προβλέπουν ε, τα εξή. Υπάρχουν και παράγοντες μετριασμού ε, στο άρθρο 23 του κανονισμού των Εγκαιρετικών και Επενδυτικών Ταμείων. Μετά τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κατά την υιοθέτηση του κανονισμού, χαίρομαι ιδιαίτερος και είμαι και προσωπικά ευγνώμων που έχουμε αυτή τη ε, δυνατότητα, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουμε ακριβώς αυτούς τους ε, παράγοντες μετριασμού. Γιατί έτσι έχουμε περιθώριο ευελιξίας, ε, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε χρόνο στα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις συστάσεις και με την απόφαση του Συμβουλίου για το επίπεδο των, της αναστολής ε, θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές και κοινωνικές ε, συνθήκες στα κράτη-μέλη, λαμβάνοντα υπόψη ιδίω το επίπεδο της ανεργίας που είναι υψηλό και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε επί της αρχής να υποβάλει πρόταση αναστολής κάτω από το μέγιστο όριο που προβλέπεται στον κανονισμό. Βάσει των προγραμμάτων που θα πληγούν από την αναστολή, η ε, λογική διάταξη είναι ότι η αναστολή θα ε, ισχύσει αναλογικά για όλα τα ε, προγράμματα και προτεραιότητε των διευθυντικών και επενδυτικών ταμείων. Όμως, ο κανονισμός προβλέπει ότι υπάρχουν ορισμένα προγράμματα και προτεραιότητε που θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή τη αναστολή, ιδίω αν πρόκειται για προγράμματα κέρια σημασία για την αντιμετώπιση των ε, δυσχερών οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων, ιδίω σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων. Να υπενθυμίσω όμως ότι η εξαίρεση ορισμένων τέτοιων προγραμμάτων από ε, τα μέτρα αναστολής δεν θα περιορίσει το συνολικό της εύρος. Επομένως, τα επίπεδα αναστολής των ε, προγραμμάτων που δεν έχουν εξαιρεθεί θα πρέπει να αυξηθούν αντιστοίχως. Αυτό ενέχει δύσκολες επιλογές ε, μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, και βεβαίω πρέπει να υπάρχει και επαρκή τεκμηρίωση γιατί ορισμένα προγράμματα κρίνονται πιο σημαντικά από άλλα. Θέλουμε να ακούσουμε και εδώ τις δικές σας απόψεις και βέβαια μετά την γνωμοδότηση που θα εκπονήσει το Κοινοβούλιο, το Σώμα των Επιτρόπων θα λάβει την ε, απόφασή του. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλια και ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Και δεν μπορώ να αποφύγω να κάνω ένα μικρό σχόλιο γιατί είμαστε νομοθέτες ε, και φυσικά σεβόμαστε τα μάλλα την ε, επιθυμία του νομοθετή αλλά εγώ δεν θυμάμαι ε, ουσιαστικά ότι ε, υπήρχε ένα είδος κύρωσης. Ε, εμείς δεν θεωρήσαμε ότι είναι θετικό το θέμα της αναστολής των κονδυλίων. Είναι ένα σκληρό μέτρο και γι' αυτό το συζητούμε. Μάλιστα είναι τυπικό σχόλιο από την πλευρά του Κοινοβουλίου αυτό. Αλλά να υπενθυμίσω στα μέλη των δύο επιτροπών ότι θα διαιρέσουμε σε δύο μέρη τη συνεδρίασή μας από εδώ και πέρα και θα ξεκινήσουμε με τους εκπροσώπους της Επιτροπής ε, Ρέτζι. Θα ήθελα να σας ζητήσω να σεβαστούμε το χρόνο, γιατί από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο για να θέσουν ερωτήσεις και οι εκπρόσωποι από τους δύο επιτροπές και για τις απαντήσεις από την Κομισιόν. Γι' αυτό προτείνω στα μέλη της Ρέτζη δύο λεπτά για τους συντονιστές για τις ερωτήσεις και τις προτάσεις τους και ένα λεπτό για το δεύτερο γύρο, αν υπάρξει. Για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη λυπάμαι, αλλά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ο συνήθως δεν μας ήταν ο χρόνος. Και μετά από τον πρώτο γύρο με τους συντονιστές. Θα δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους να απαντήσουν και θα περάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο γύρο. Θα ξεκινήσω τώρα με τους συντονιστές με τη σειρά. Να το κόλλω δύο λεπτά. Ο καθένας, καταρχήν ο κύριος Λαμπέρτ Ρόι από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ξεκινάμε αυτό το διαρθωτικό διάλογο. Εγώ ήμουν στις διαπραγματεύσεις πριν 4-5 χρόνια και θυμάμαι όλα όσα συζητήθηκαν εκεί. Και να είμαι πιο συγκεκριμένος, όταν μιλήσαμε για αυτές τις δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 23, αυτό ήταν ε, μια έσχατη λύση. Δεν είναι κάτι γραφειοκρατικό, δεν είναι ε, κάτι ρομποτικό αυτόματο όπως είπε η Κομισιόν, είναι μια έξυπνη, μια ευφύης προσέγγιση. Ή Επιτροπή σας είναι μια πολιτική επιτροπή, το είπατε, είναι σαφές αυτό. Αλλάξατε την πρόταση περιεγωγής, γιατί υπήρχε λόγος να μην παρουσιαστεί ε, κάτι που δεν θα ήταν λογικό και ακριβώς αυτό διακυβεύεται σε αυτό τον διαρθρωτικό διάλογο. Μπορώ να σας πω ότι αν δούμε το πώς το διατυπώσαμε όλο αυτό το θέμα, δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία βομβαρδισμού. Μπορείτε να πείτε δεν έχει να κάνει με τις πληρωμές. Ναι, ποτέ δεν ήταν ο σκοπός να φύγει τις πληρωμές, αλλά μιλάμε για τις ε, νέες αναλήψεις υποχρεώσεων από πρώτη πρώτου του χρόνου. Και ε, αν δείτε τι γίνεται με την Πορτογαλία που τα επενδυτικά χρήματα έρχονται από την Ευρώπη, πραγματικά ε, ουσιαστικά πλήττεται την καρδιά της χώρας, ε, πλήττεται το εκπαιδευτικό σύστημα, το ενεργειακό, τους αγρότες. Έτσι λοιπόν Λοιπόν, ποιο ρόλο έχει αυτός ο διαρθρωμένος διάλογος, να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα να βρούμε κάτι άλλο. Εγώ τώρα είμαι η συγητής για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Και τι σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει τα χρήματα από τα ταμεία να υποστηρίζουν τις χώρες, ιδίως την Ισπανία και την Πορτογαλία, να τα πάνε καλύτερα και να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις εδώ. Δεν μιλάμε για χρήματα και περικοπές, αλλά για ευφυΐα. Και τελευταία πρόταση, καλό την Επιτροπή σας και θέλω μια απάντηση σε αυτό, να παρουσιάσει μία ουσιαστικά πρόταση που να είναι σωστή. Δεν τιμωρήσετε το κράτος, αλλά τώρα θέλετε να πλήξετε εδώ τους δικαιούχους. Ευχαριστώ κύριε Βανίστεν Ρόι. Πολύ καλή αρχή ε, για το διάλογο. Κύριε Σκοτσουλίνο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Εμείς ε, θεωρούμε το μέτρο αυτό παράλογο και όχι και ιδιαίτερα ευφυές όπως ε, υπόθηκε. Και μάλιστα ε, είμαστε ή μιας εποχής πολιτικής. Όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση, ο τριμερής διάλογος υπό το αίτημα της Κομισιόν μαζί ζήτησε αυτή τη δέσμευση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος ε, Φανής Τελερόη. Και ακριβώς ε, εδώ βλέπουμε την πολιτική της παλιάς Κομισιόν. Εμείς πάντοτε είμαστε αντίθετοι πέρα από τους πολιτικούς προσανατολισμούς. Η Επιτροπή Ρέτζι αντιτίθεται πάντα ε, σε ένα τέτοιο σκεπτικό γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Ε, μάλιστα είναι κάτι παράλογο και από τη σκοπιά της οικονομικής διακυβέρνησης γιατί διακόπτει ένα, δημόσιο, ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων όταν παρεμβαίνει επί των πληρωμών, γιατί ζημιώνει σοβαρά την επιτυχία των ιδίων των προγραμμάτων όταν ε, ουσιαστικά ε, μιλάμε για τις αναλήψεις υποχρεώσεων γιατί αναστέλει τον προγραμματισμό και τις επιλογές ε, της χώρας αυτής και παράγει ουσιαστικά συνέπειες, έχει συνέπειες για την τοπική κοινότητα όπως πολύ σωστά υπενθυμίσαμε εδώ. Επομένως, εμείς θέλουμε να πούμε το εξή. Πάντοτε ευχόμαστε αυτό το μετρό να μην λαμβάνεται υπόψη, να είναι ουσιαστικά κάτι έσχατο. Και πάντοτε έτσι το ερμηνεύαμε ως Επιτροπή Ρέτσι. Τώρα, παραδόξως, και αυτή είναι η ερώτηση που θα θέτουμε, γίνεται η πρώτη λύση. Γιατί εσείς ως Επιτροπή, και καλά κάνετε κατά την άποψή μου, να εισαγάγετε ένα μηχανισμό επιβολής προστήμων για τις δύο χώρες, αλλά την πολιτική συνοχή στη μετατρέπεται ακριβώς σε μια πολιτική προστήμων. Πριν λοιπόν να μπούμε στην ουσία που θα το κάνουμε σε αυτό το διαρθρωτικό διάλογο, στο διάλογο, θέλουμε να καταλάβουμε και τα νομικά επιχειρήματα τη απόφασή σας, τη νομική βάση και τι ακριβώς θα κάνετε τη στιγμή που θα προχωρήσετε στην υιοθέτηση της ιδέας της αναστολής της χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Τόμασίτς από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Το ECR συμφωνεί ότι οποιαδήποτε απόφαση που συνδέεται με την αναστόλη διαθετικών και επιθετικών ταμείων θα πρέπει να έχει τύχη ε, χρηστή εξέταση, να είναι πλήρω ε, τεκμηριωμένη και να είναι πραγματικά έσχατη λύση. Υπάρχει ισχύ σε αυτέ τι κυρώσει, ε, όμω είναι αδιαφεσβήτητο ότι η αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήττεται κάθε φορά που κινητοποιούνται και δεν επιβάλλονται. Ε, Βεβαίω και κατανοούμε και συμπάσχουμε με του Ισπανού και Πορτογάλου που όπω και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Ακόμα και ένα συμβολικό πρόστιμο ε, θα είχε θεωρηθεί από εκείνου ω μια ε, πολύ βαριά τιμωρία. Όμω αναγνωρίζουμε ότι ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον είναι απαραίτητη προπόθεση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ε, και επιχειρηματικότητα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα κατάλληλο χρηματοδοτικό μέσο και να τηρούνται οι κανόνες του. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βαν Μιλτεμπουργκ από την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίζουμε και τους δύο επιτρόπους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επειδή διάβασα στο Πολίτικο την περασμένη Παρασκευή ένα αρθράκι ε, που παρέπεμπε και στη δική σας ενημέρωση, στο δικό σας briefing και το ε, συνιστώ σε όλους, ήταν πολύ σαφές. Λέτε ότι υπάρχει νομική υποχρέωση σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, άρθρο 23, παράγραφος 9, Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση κινητοκίνησης αυτής της διαδικασίας όταν πληρούνται αυτές τις προϋποθέσεις. Πολύ λυπούμεθα που πρέπει να το κάνουμε. Παρά τις μεγάλες, τεράστιες θα έλεγα προσπάθειες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, τώρα βρισκόμαστε ενώπιν αυτής της κατάστασης. Υπάρχει δήλωση του Συμβουλίου που λέει ότι δεν, υπήρξε, ε, δεν υπήρξαν επιτυχείς αποτελεσματικές ενέργειες υπό τη δικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και όταν λέμε ότι συνδέουμε τις επενδύσεις υπό, το, ε, υπό τα ταμεία ΕΖΗ, πρέπει να τα συνδέσουμε, λέμε, με μια χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Επομένως, μπορούμε να πούμε ναι, κρίμα. Όμως υπάρχουν κανόνες και θα πρέπει όλοι να τους στηρούμε. Ιδάλω δεν θα υπάρχει οικονομική διακυβέρνηση. Βεβαίω, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει ε, προσαρμοσμένε ε, στην πραγματικότητα λύσει και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, μείωση τη φτώχεια και ούτω καθεξής. Αν δείτε το παράρτημα 3 και το άρθρο 23 ε, του κανονισμού κοινών διατάξεων υπάρχει κάτι που σχετίζεται με το πεδίο εφαρμογή και τα επίπεδα της αναστολής ε, των, ε, αναλήψεων υποχρεώσεων. Έχετε μια πρώτη εκτίμηση σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, το εύρος της αναστολής. Ήδη τον Ιούλιο ε, υπήρξε μια επιστολή που ανέφερε όλα τα προγράμματα, όμως θα ήθελα και τώρα να μου πείτε ποιο είναι το επίπεδο. Πότε να περιμένουμε την πρόταση, εντός ενός μήνα και θα ξαναέρθετε εδώ στο Κοινοβούλιο να μας τα εξηγήσετε μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ομαζέ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Στο άρθρο 23 προβλέπεται ένας διαθεωμένος διάλογος και αυτό γιατί όλοι φοβούμεθα μήπως φτάσουμε στα χειρότερα. Δυστυχώς εδώ φτάσαμε. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν το μοναδικό θεσμικό όργανο που πολέμησε μέχρι την τελευταία στιγμή, πάλεψε για την εισαγωγή αυτών των διατάξεων και υπάρχει μια συμβατότητα σε σχέση με αυτό που αναφέρει αφενός ε, το Συμβούλιο να μην επιβάλλει ε, πρόστιμα και από την άλλη το Κοινοβούλιο που έχει καταπολεμήσει αυτή την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα να λέει ότι είναι υπέρ τη αναστολή των ταμείων που για μας είναι μια άδικη, παράλογη και επικίνδυνη κύρωση. Αδική γιατί ε, πλήττονται οι περιφέρειες. Αυτές είναι που θα πληρώσουν το βαρύ ε, τίμημα των ε, δημοσιονομικών πολιτικών που είναι εντελώς εκτός της εμβέλειάς τους. Είναι παράλογες γιατί δεν συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας στις περιφέρειες που είναι οι πλέον ευάλωτες όπως είναι αυτές στις περιφέρειες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Και τέλος είναι και επικίνδυνες αυτές οι κυρώσεις για το ευρωπαϊκό εγχείρημα γιατί η πολιτική συνοχής δεν είναι μία μεταβλητή προσαρμογή ε, των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ούτε πρέπει να ε, τεθεί στην υπηρεσία των ε, κρατών που θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το επίβλεπε και ε, τιμώρησε. Εάν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτή την οδό, πραγματικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν θα μπορεί κανείς να το περασπιστεί πλέον. Θέλουμε κάτι τέτοιο μετά το Brexit. Αυτό το ερώτημα έχω εγώ να θέσω. Και κάτι ακόμα, νομίζω ότι καλό θα ήταν να επιβάλλουμε κυρώσει στα κράτη που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε των Πρεσίμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους κυρίους επιτρόπους εδώ. Θέλω να σας πω ότι και οι πράσινοι είναι κατά της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Θεωρούμε ότι η αναστολή αυτών των ε, ταμείων για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι κάτι εντελώς αντιπαραγωγικό. Αντιπαραγωγικό μέτρο γιατί θα θίξει περιοχές, πόλεις, και ε, αυτό επειδή έχουν γίνει λάθη σε εθνικό επίπεδο και επίση είναι μια διπλή τιμωρία για όσου είναι σε πιο ευάλωτη κατάσταση και για κοινότητες που για χρόνια χρειάστηκε να αγωνιστούν για την ύπαρξή τους αλλά κυρίως είναι αντιπαραγωγικό γιατί μια αναστολή αυτών των κονδυλίων θα συνεχίσει να διαιρεί την Ευρώπη και να καταστρέφει την ελληνική μεταξύ των κρατών μελών. Ιδίω αυτούς τους καιρούς μετά το Brexit ε, απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση, μεγαλύτερες επενδύσεις και όχι αναστολή των κονδυλίων. Αυτό θα ήταν εντελώς λάθος μήνυμα που θα προκαλούσε μεγάλη ζημία. Οι ερωτήσει μου, γιατί εσείς κυρία Κρέτσου αναφερθήκατε σε κάποιους παράγοντες μετριασμού και για αυτού έχει αγωνιστεί ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Ποιοι οι παράγοντε μετριασμού και σε ποιο βαθμό θα εφαρμοστούν ε, προκειμένου να υπάρχει μείωση του αντικτύπου της αναστολής. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι το 50%. Ποιες πληροφορίες μπορείτε να μας δώσετε για αυτούς τους παράγοντες μετριασμού εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ενημερωθεί ορθά το Κοινοβούλιο για να μπορέσει να ελοποιήσει αυτό το διάλογο. Και επίσης ε, για ποια δημοσιονομικά ποσά μιλάμε. Αυτός ο διαρθρωτικός διάλογος θα πρέπει να έχει ένα δυναμικό πολύ μεγαλύτερο ε, πέρα από το να γίνεται στο πλαίσιο μιας ακρέωση. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εγκρίνει ένα ψήφισμα και να ψηφίσει για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, το κίνημα πέντε αστέρων κρίνει τις αρχές της μακροοικονομικότητας. Είμαστε εντελώς ε, αντίθετοι ε, γιατί υποσκάπτει ουσιαστικά τις ε, ε αρχές και βλέπουμε να αυξάνεται ε, από την κεντρική κυβέρνηση. Ε, τελικά αυξάνονται τα λάθη και σήμερα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το άρθρο 23 έναντι δύο χωρών που έχουν λάβει δρακόντια μέτρα λιτότητας ε, και η πολιτική συνοχής μπορεί ε, να ε, βελτιωθεί αλλά παραμένει το κύριο εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, το να εμπλέκουμε το Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και της ενεργοποίησης του άρθρου 23 είναι κάτι απαραίτητο για να έχουμε μια αναδιανομητική πολιτική για να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Πραγματικά ε, μας απογοητεύει ότι εφαρμόζονται κάποια τέτοια κριτήρια για τα επιχειρησιακά προγράμματα των δύο χωρών. Έτσι θέλετε να καταπολεμήσετε τον ευρωσκεπτικισμό που τόσο σας ανησυχεί. Έχουμε δύο χώρες σε δύσκολη θέση και εσείς τις τιμωρείτε. Ακόμη περισσότερο η έννοια της ελληνικής υπάρχει στις ευρωπαϊκές συνθήκες, όμως ίσως να το ξέχασε η Κομισιόν. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι και ο ίδιος ο Υπουργός τη πορτογαλία ε, είπε ε, ότι είναι τιμωρητική η εφαρμογή ε, της αναστολής των αλήψεων υποχρεώσεων δεν θα ήταν κάτι που θα κατανοούσε ο πληθυσμός και σίγουρα θα έπλητε κάποια ε, project σε περιφερειακό επίπεδο. Μπορεί η Κομισιόν να μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για την κοινωνικονομική κατάσταση των δύο χωρών. Ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος της αναστολής. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση. Δεν ακούσαμε αυτά τα στοιχεία σήμερα. Δεύτερον, η παράγραφος 16 του ιδίου άρθρου λέει ότι η Κομισιόν το 2017 θα πρέπει να επανεξετάσει το σημερινό άρθρο, να παρουσιάσει μια έκθεση και να προτείνει, να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση. Η οικονομική ανάπτυξη είναι χειρότερη αυτή του 2013, έτσι λοιπόν οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. I don't see Mr. Δεν βλέπω εδώ τον ε, κύριο Μπριουά. Επομένως, αυτές ήταν οι ερωτήσεις ε, από τους συντονιστές της Επιτροπής Ρέτζη. Κυρία Κατάινεν, κυρία Κρέτσου, έχετε τώρα το λόγο για να απαντήσετε. Σας παρακαλώ μέσα σε 4-5 λεπτά, αν είναι δυνατόν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε βουλευτές για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ανησυχίες σας όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια και η Κρέτσου θα μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν θέλω να υπογραμμίσω το εξή. Η Κομισιόν έχει νομική υποχρέωση να αναλάβει δράση. Αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά έχουμε νομική υποχρέωση. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεύτερον, η αναστολή, η μερική αναστολή δεν είναι κύρωση. Για δύο λόγους. Καταρχήν, δεν θίγει τις πληρωμές. Και επίσης, επειδή οι κυβερνήσεις ε, μπορούν να αποφύγουν μόνιμες απώλειες, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω παρά το να γίνουν σεβαστές ε, οι αναλήψει υποχρεώσεων. Έτσι λοιπόν, οι δύο κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί στα άλλα κράτη-μέλη και στους πολίτες τους ε, να ακολουθήσουν τη δημοσιονομική οδό. Δεν έχουν δεχτεί στο Συμβούλιο Κοφίν. Και όταν θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους δεν θα χαθεί ούτε ένα σέντ. Νομίζω ότι κανένας σε αυτή την αίθουσα δεν θα πίστευε ότι αυτές οι δύο κυβερνήσεις ε, ε, δεν θα κρατήσουν τις υποσχέσεις τους στους πολίτες και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να προκρίνω τη μελλοντική απόφαση της Κομισιόν, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που αποφασίσουμε μερική αναστολή, Έχουμε σημαντικό ποσό πληρωμών και εναπομείνασες αναλήψεις υποχρεώσεων για τις δύο χώρες. Και μάλιστα πολλά περισσότερα από όσα έχουν κατορθώσει να απορροφήσουν οι δύο χώρες σε αυτή την προγραμματική περίοδο μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν ούτε ένα και μόνο έργο δεν θα τέθει σε κίνδυνο, ούτε ένα έργο. Και το τελικό μου σχόλιο έχει να κάνει με το εξή. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι σαφές για όλους, αλλά ο λόγος που έχουμε την αιρεσιμότητα στα διευθυντικά ταμεία είναι κάτι πολύ λογικό. Έχουμε εξάντε αιρεσιμότητα και έχουμε και εξπόστ αιρεσιμότητα. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι όταν ε, χρησιμοποιούμε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα χρήματα πράγματι δημιουργούν πρόσθετη αξία και χρησιμοποιούνται όπως πρέπει οι συνομοθέτες στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθώς έχουν τονίσει ότι αν η αν το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό, το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Αντίθετα, το χρήματα του φορολογουμένου, αντί αυτού μάλλον θα χαθούν τα χρήματα του φορολογουμένου. Γι' αυτό η εξάντη και εξπόστερη σημότητα είναι πολύ σημαντική προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα τα χρήματα του φορολογούμενου. Αλλά η Επίτροπος Κρέτσου θα συνεχίσει. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω στη μετρική μου. Μάλιστα. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τις απόψεις τις οποίες έχετε εκφράσει εδώ σήμερα. Είμαι πεπισμένη και εγώ ότι πρόκειται για ένα μέτρο έσχατης λύσης, όπως ανέφερε ο κ. Βανής στον Ραγιακό Τσολίνο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα όσα εξετάζουμε σήμερα δεν αποτελούν συνέπεια της αξιοποίησης, του τρόπου αξιοποίησης των ταμείων από ε, τα κράτη-μέλη, αλλά είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων του Συμβουλίου και που απορρέουν με τη σειρά τους από τον κανονισμό Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ε, ακριβώς ε, που προβλέπουν τις διατάξεις ε, που διέπουν τα επενδυτικά και διευθυντικά ταμεία. Γι' αυτό θεωρείται από το Συμβούλιο ότι δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα για τα έτη 14 και 15 στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος υπό το άρθρο 23 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να προτείνει στο Συμβούλιο την αναστολή τμήματος των αναλήψεων υποχρεώσεων ε, για αυτέ τις χώρες για την επόμενη χρονιά. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για αναλήψεις υποχρεώσεων και όχι πληρωμών. Οι πληρωμές θα γίνουν. Επιπλέον, συμφωνώ ε, και, και εγώ στηρίζω και θαυμάζω τις δύο αυτές χώρες και γνωρίζετε ότι και εγώ αγωνίζομαι ε, για τον ε, μετριασμό και την εξομάλυνση των ανισορροπιών. Ε, την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκα τη Μαδέιρα που είχε πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι και με μεγάλη μου χαρά μπορούμε να στηρίξουμε την περιφέρεια αυτή με το Ταμείο Λιλεγγύης. Ξέρετε ότι και εγώ δεν είμαι σε εύκολη θέση όταν πρέπει να πω ότι θα πρέπει να αναστείλουμε τμήμα των πιστώσεων για το 2017. Αλλά έτσι προβλέπει η νομοθεσία μας. Άκουσα και τις δύο κυβερνήσεις που είπαν ότι στις 15 Οκτωβρίου θα υποβάλουν έκθεση που θα καταδεικνύει ακριβώς ε, τα σημαντικά βήματα που θα πραγματοποιήσουν για το ε, Σύμφωνο Σταθερότητας για τα στοιχεία που ζητήσατε. Από το 2014 2020, 26 δις θα λάβει η Πορτογαλία. Για την Ισπανία, στο πλαίσιο των Ταμείων Συνοχής, 38 δισεκατομμύρια ευρώ θα λάβει. Για το 2014-2016, σας έδειξα πριν αυτό το γράφημα, για την περίοδο 2014-2016 λοιπόν, 8,2 δις αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν ήδη διχετευτεί, 1,5 δις έχει δαπανίσει μέχρι τώρα η Πορτογαλία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα στοιχεία επαρκούν για να δείξουν αυτό που ανέφερε ο Γύρκη, ότι υπάρχουν κονδύλια στη διάθεση των χωρών αυτών μέχρι το 2020 θα είναι μικρό το τμήμα ε, που θα ανασταλεί, εάν ανασταλεί τελικά. Το λέω και πάλι, αυτές οι δύο χώρες έχουν ε, δαπανίσει όχι και πολύ μεγάλο ποσό για την περίοδο 2014-2016. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτές τις δύο χώρες, ε, για να αξιοποιήσουν τα ταμεία προς όφελος των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο έχει αποφασίσει το Συμβούλιο ε, να αναβαθμίσει τα δημοσιονομικά μέτρα για να υπάρξει συμμόρφωση με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Τώρα, για τους ε, παράγοντες μετριασμού. Η κυρία Βάνα, αν δεν κάνω λάθος, ε, έθεσε ένα ερώτημα που αφορούσε το ποσοστό ανεργίας που είναι πολύ υψηλό και στις δύο αυτές χώρες τα επίπεδα αναστολών ενδέχεται να μειωθούν σημαντικά εάν λάβουμε υπόψη και το ποσοστό ανεργίας. Αν είναι 8% μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί η αναστολή να περιοριστεί κατά 50%. Και είμαστε βέβαιοι ότι αν συζητήσουμε αυτή την αναστολή, θα λάβουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες που αναφέρονται στον κανονισμό. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις απαντήσεις. Έχουμε τέσσερις ακόμη ομιλητές. Έχω ένα κατάλογο. Επιθυμεί άλλος να πάρει το λόγο. Κύριος Μποστινάρου, πέμπτος, μάλιστα. Κύριε Βαλίνα. Ακτή ομιλήτρια, έξι άτομα λοιπόν. Κύριε Ρούας. Είστε ο πρώτος. Θα δώσω λοιπόν το λόγο σε επόμενους ομιλητές από την Επιτροπή Ρέτζι, Ένα λεπτό παρακαλώ. Λίγο παραπάνω ίσως, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ προέρχομαι από τις δύο χώρες και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα Καταρχήν ε, για το θέμα της μέγιστης ε, ευελιξίας ε, των κανόνων, το οικονομικό πλαίσιο των δύο χωρών και τη διαδρομή τους και τα αιτήματα των κυβερνήσεων πρέπει να λάβουμε υπόψη και επίσης το τα αρνητικά αποτελέσματα που έχει αυτή η συζήτηση στους πολίτες αυτής της χώρας αλλά και στις επενδύσεις. Εγώ θα ήθελα να πω από, τη συνθήκη, από την σύσταση της 27 ε, Ιουνίου και την απόφαση ε, του Συμβουλίου τι συνέβη, δηλαδή ότι ίσχυσε για να μην επιβληθούν τα πρόστιμα δεν ισχύει και για το θέμα της αναστολής ε, θα ήταν παράλογο να μην γίνει κάτι τέτοιο πώς θα εξηγούσαμε στους πολίτες μας αυτό το βαθύ άδικο μετά από τόσες θυσίες που έκαναν για να επαναφέρουν τη χώρα στη σωστή οδό και μιλώ για τις θυσίες της Πορτογαλίας, των πολιτών, των επιχειρήσεων και Πώς είναι δυνατόν λοιπόν τη στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προωθήσει τις επενδύσεις, ε, να ε, επιβάλλει τέτοιες κυρώσεις που δεν ευνοούν την ανάπτυξη οι κύριοι επίτροποι ξέρουν ε, ότι το 2014-2016 το 12% των επενδύσεων στην Πορτογαλία προήρθε από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και ξέρετε αν ληφθεί αυτή η απόφαση πόσο αρνητικές επιπτώσεις θα είχε ε, στις ε, δύο χώρες θα ήθελα να κλείσω να πω το εξής. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των διάφορων οικονομικών συνθήκων ε, βάσει του άρθρου 23 ε, και να δούμε ότι το μόνο που μπορούμε να εξαγάγουμε ως συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να επιβληθεί αυτή η αναστολή στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Κυρία Ροντρίγκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η αναστολή των ταμείων για την Πορτογαλία είναι άδικη απέναντι στις δημοσιονομικές προσπάθειες που κάνει η Πορτογαλία, είναι άδικη και μπροστά στις διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη αναλυφθεί. Έχουμε φτάσει στις δεσμεύσει μα σύμφωνα με το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα και το Σύμφωνο σταθερότητα. Και είναι άδικο γιατί η κυβέρνηση τη πορτογαλία του 2016 θα φτάσει σε ένα έλλειμμα κάτω του 3%. Είναι αντιπαραγωγικό και θα έχει άμεση αρνητική ανάπτυξη στην οικονομία, στι επενδύσει, στην καταπολέμηση τη ανεργίας και τη φτώχεια και δεν είναι συνεκτικό με την απόφαση που ελήφθη από την Κομισιόν και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο να μην επιβληθούν τα πρόστιμα. Δεν θεωρώ ότι η αναστολή ε, των ε, κονδυλίων ε, είναι ουσιαστικά κάτι που πρέπει να γίνει. Ξέρετε πόσο αντίκτυπο έχουν αυτά τα κονδύλια και ξέρετε πώς είναι ο σκεπτικισμός από την πλευρά των πολιτών που ουσιαστικά έζησαν τέσσερα χρόνια σκληρής κρίσης και να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος ουσιαστικά θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στο τι υπόθηκε σε αυτό το άρθρο που, στον οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφο την Παρασκευή. Ευχαριστώ. Κύριο ε, Βαλκάρ Σελσίσο, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Αυτός ε, ο διαρθρωμένο διάλογος ελπίζουμε να μην ε, γίνει ένα στήριο διάλογος γι' αυτό γιατί ακούγοντα του εκπροσώπου τη Κομισιόν του οποίου φυσικά σέβομαι Συνειδητοποιώ ότι εδώ δεν γίνεται τίποτα, ε, μας έρχεται και μας λέτε, κοιτάξτε μην ανησυχείτε, παίρνουμε κάποια μέτρα γιατί το λένε οι κανονισμοί και πολιτικά δεν υπάρχουν συνέπειες ε, ε, εκτός από κάποιες οικονομικές. Όμως αν είναι έτσι τι κάνουμε όλο αυτό τον καιρό. Γιατί χάνουμε αυτό το χρόνο εκεί, γιατί να προκαλούμε γενικευμένο θυμό όπως ε, και άλλοι που πήραν το λόγο πριν και εγώ είμαι εντελώ αντίθετος σε αυτό το μέτρα γιατί είναι άδικα, δεν είναι κατάλληλα και δεν είναι αναλογικά το έκανε Πορτογαλία, το έκανε και η Ισπανία. Ε, μισό εκατομμύριο θέσει εργασία κάθε χρόνο στην Ισπανία και τελικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα κράτη-μέλη που αναπτύσσονται περισσότερο. Και τώρα πρέπει, επειδή δεν έκανε τι ασκήσει στο σπίτι, πρέπει να την τιμωρήσουμε. Ε, Δυστυχώ πρέπει να δούμε ότι τέτοιες πράξεις καταστρέφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταστρέφουν την δυνατότητα να έχουμε ένα ευίωνο μέλλον. Θα πρέπει να είμαστε πιο δίκαιοι και να μην τροφοδετούμε την έλλειψη σύγκλησης. Η πολιτική συνοχής βοηθά στη σύγκληση και να αποφύγουμε με κάθε μέσο να δημιουργείται βεβαιότητα κυρίως ε, σε όσους ε, έχουν επενδύσεις ε, σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές με περιφερειακή πιστοποίηση γιατί από τη στιγμή αυτή αυτή η αβεβαιότητα μπορεί να προκαλέσει μια ολική παράλυση στην ανάπτυξη των περιφερειών αλλά και των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βγασό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι άχρηστη όλη αυτή η άσκηση, είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο με ένα τρόπο που μου φαίνεται τόσο ξεκάθαρος που δεν μπορείτε να προσπεθείτε ότι δεν το καταλαβαίνετε, σας λέει ότι ε, δεν κατανοεί ότι να υπάρχουν οι για να εφαρμοστεί το άρθρο 23. Εμεί δεν θεωρούμε ότι πληρούνται οι προποθέσει. Οι δύο χώρε έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειε και συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τεράστιε προσπάθειε και επομένω να τις τιμωρήσουμε αυτή τη στιγμή επιλέγοντας ε, ε, ουσιαστικά κάτι που παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητα, ε, παραβιάζει την αρχή ότι όταν δημιουργείται ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις επενδύσεις ε, πρέπει να σεβόμαστε τι αρχέ ε, και ε, ε, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής είναι σε επενδύσεις που είναι βέβαιες και δημιουργούν ε, προοπτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας. Όλα αυτά θα έπρεπε να σας κάνουν να σκεφτείτε ότι είτε αστευόμασταν ε, όταν ε, ε, με αυτό το διευρωμένο διάλογο ή εσείς θα πρέπει να επανέλθετε στο Συμβουλίο και να πείτε ότι θεωρείτε ότι δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η Επιτροπή δεν είναι εκτελεστικό όργανο, αλλά εκπροσωπεί όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Έτσι λοιπόν, εμείς σας λέμε ξεκάθαρα θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί αυτό το άρθρο. Πρέπει να σας διακόψω σου. ο ομιλητή, η κυρία Βαλίνα, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Καλησπέρα σα. Εγώ νομίζω ότι η αναστολή των πληρωμών είναι κάτι ανήθικο και δεν είναι συνεκτικό ούτε νόμιμο και είναι ανήθικο δεν μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερες περικοπές στα δικαιώματα των πολιτών ε, και δεν είναι συνεκτική γιατί τα ταμεία θέλουν να εγγυηθούν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική συνοχή ενώ εδώ θα έχουμε τον τελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το άμεσο αποτέλεσμα που θα πετύχουμε θα είναι ε, ε, απόλυτη αστάθεια και παράνομα γιατί όπως λέει το άρθρο 23 στο σημείο 11, θα πρέπει να σέβονται την αναλογικότητα και την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και να ληφθούν υπόψη και οικονομική καταστάσεις και το επίπεδο της ανεργίας. Και ξέρετε, πρέπει να το δείτε και αυτό για την Ισπανία. Εδώ ε, ουσιαστικά τι θέλετε, μας λέτε ότι θέλετε να εφαρμόσετε την αρχή της ισότητας. Δεν ξέρω και τον σύμφωνα με το ΙΦΟΠ. Ε, ε, όλες οι χώρες και οι σε χώρε από τη στιγμή που θετήθηκαν τα κριτήρια του Μάστερ δεν έχουν σεβαστεί του κανόνε περί ελλείμματο. 14 φορέ, ε, λέει το Ινστιτούτο έχει γίνει. Πού είναι λοιπόν η αρχή τη μεταχείριση, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Είναι μήπω ε, κράτη που έχουν λιγότερα δικαιώματα από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου, για ένα λεπτό παρακαλώ. Μάλιστα, ένα λεπτό θα μιλήσω μόνο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, δεν ε, θα σας καλέσω να διαβάσετε και πάλι ε, τις κατηγορίες που υπάρχουν για την, αυτό το δόγμα του 3%. Θα ήταν βέβαια πολύ ενδιαφέρον αυτό το ανάγνωσμα, όμως ας αφήσουμε στην άκρη το Στίγκλης. Εσείς προτείνετε πρώτα και πόλα πολιτικά και ηθικά ε, εσφαλμένες ε, κυρώσεις για δύο χώρες που ήταν αυτές που επλήγησαν μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την ε, κρίση και θέλετε να συνεχίσετε τη λιτότητα. Δεύτερον, τιμωρείτε τις περιφέρειες βάσει πολιτικών που υιοθετήθηκαν από εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Και και η Επιτροπή ε, Ρέτζι αλλά και η Επιτροπή των Περιφερειών πάντα καταδικάζουν ακριβώς αυτή τη στάση. Ποιο θα είναι το μέλλον της πολιτικής συνοχής και για το σημερινό πολιτισμικό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικέ οι επιπτώσει αυτών των κυρώσεων. Και σα καλώ να ρίξετε μια ματιά και στον σορευτικό αντίκτυπο αυτών των μέτρων για τις χώρες που υλοποιούν τη νέα πολιτική συνοχή. Να θυμάστε και την περίπτωση της Ρουμανίας, όπου ανεστάλησαν έξι επιχειρησιακά προγράμματα για μάλλον ασαφείς λόγους. Ε, κατηγορούμε την άνοδο του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού, αλλά ας κοιτάξουμε και λίγο τι συμβαίνει ε, στο σπίτι μας αν θέλετε. Ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2019 αν θέλετε να δείτε τι θα συμβεί, σκεφτείτε τι κάνετε ακριβώς σήμερα. Γιατί αυτό το κοινοβούλιο είτε θα στηρίξει την Ένωση είτε θα την μπλοκάρει. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φερνάντες. Λυπάμαι, δεν ήξερα ότι υπάρχει αντικατάσταση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα έχω να κάνω μια πολύ δύσκολη παρέμβαση και είναι πολύ δύσκολη γιατί πρέπει να περασπίσω τους ε, Ισπανούς πολίτες από μια κυβέρνηση που δεν έκανε όσο θα έπρεπε για ε, να καταπολεμήσει το έλμα και ουσιαστικά ενέκρινε ένα φορολογικό σύστημα που ευνόησε τα νότερα στρώματα. Θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να αναλύσει καλά την απόφασή της και να λογιστοποιήσει οποιαδήποτε εμπλοκή των διαφορετικών ταμείων. Αν η Κομισιόν ε, δεν μπορεί να αποφύγει εντελώ την ευθύνη σας, παρακαλώ να μας εξηγήσετε με σαφήνεια ποια είναι η μεθοδολογία, ποιο είναι το σύστημα πώς εσείς θα υπολογίσετε αυτή την αναστολή των ε, διαφορετικών ταμείων, γιατί θα πρέπει να ε, έχουμε όλα τα στοιχεία προκειμένου και αυτό το Κοινοβούλιο να πιέσει το Συμβούλιο για να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση σε αυτό το θέμα. Ποια απάντηση έχει η Κομισιόν ε, για ανήθικα ε, και παράνομα το όπως έγιναν στην Ουγγαρία πριν λίγους, ε, πριν μήνες ε, ουσιαστικά δεν μπορούμε την Ευρώπη να την συρρυκνώνουμε και να μιλάμε μόνο για ελλείμματα η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από αυτούς τους αυτόματους κανόνες γιατί πρέπει να προσφέρουμε κάποια ελπίδα στους πολίτες θα θέλαμε να μας προσφέρετε έναν ορίζοντα. Σκεφτείτε ότι το ευρωπαϊκό ε, σχέδιο, το ευρωπαϊκό όραμα είναι στα χέρια σας. Δώστε μας μια ελπίδα να σώσουμε την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ήταν η τελευταία παρέμβαση από την Επιτροπή Ρέτζη. Παρακαλώ κύριε Επίτροπη, θέλετε τώρα το λόγο να αντιδράσετε. Ευχαριστώ πολύ. Αντικατέστησε το μέλος από την Επιτροπή Ρέτζη, λέει η Πρόεδρος. Λυπάμαι είναι κάτι το οποίο ε, έχουμε διαπραγματευτεί εγώ με τον ε, πρόεδρο της ΕΙΚΟΝ και ο κύριος αντικατέστησε έναν από τους εκπροσώπους ε, της Επιτροπής Ρέτζη και αξιοποίησε αυτό τον χρόνο ακριβώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Κύριε Επίτροπη, θέλετε να πάρετε τον λόγο. Παρακαλώ, ο κύριος Κατάινεν. Τρία-τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ε, τέθη το ζήτημα της ευελιξίας. Όπως βλέπετε, όπου η Επιτροπή είχε μια επιλογή, όπου υπήρχε περιθώριο ευελιξίας, εμείς εφαρμόσαμε το μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας και με τις δύο αυτές χώρες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν έλαβαν πρόστιμο. Όμως υπήρχε νομική υποχρέωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνουμε την μερική αναστολή των ε, πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων. Είναι μια διαφορετική νομοθετική πράξη. Δεν ξέρω αν, το έχετε καταλάβει όλοι. Ακριβώς αυτή τη στιγμή όπου οι δύο κυβερνήσεις υποβάλλουν σχέδια προπολογισμού που συμμορφούνται με τις, ε, ε, με τις προοπτικές που έχουν αποδεχθεί οι δύο κυβερνήσεις. Η Επιτροπή λοιπόν εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή θα άρει ε, την αναστολή. Επομένως αναπόκειται στα κράτη-μέλη. Ούτε ένα σεντ δεν θα χαθεί, αρκεί οι κυβερνήσεις αυτές να πράξουν τα όσα έχουν ήδη υποσχεθεί ενώπιον των πολιτών τους και ενώπιον άλλων κρατών μελών. Εγώ τουλάχιστον είμαι βαθιά πεπισμένο ότι οι δύο κυβερνήσει θα κάνουν αυτό που έχουν υποσχεθεί επειδή το έχουν υποσχεθεί και κατανοούν τη σοβαρότητα τη κατάσταση και δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας τους. Επομένως, εναπόκειται στα κράτη-μέλη αυτή η υπόθεση. Κάποιος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τιμωρήσει τις περιφέρειες, γιατί οι κυβερνήσεις δεν ε, παίζουν βάσει κανόνων. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν ευμερούσες περιφέρειες ε, όταν δεν πηγαίνουν καλά οι κυβερνήσεις. Και το αντίθετο βέβαια. Μόνο μία είναι η οικονομία. Επομένω, πρέπει να έχουμε και μια ισχυρή εθνική οικονομία και ισχυρές περιφερειακές οικονομίες. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Γι' αυτό και υπάρχει μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Κάτι επί το οποίο εύκολα μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι κανέναν δεν συμφέρει να χαθεί έστω ένα σέντ από αυτά τα χρήματα. Και είναι όχι μόνο εφικτό, αλλά είναι και πολύ πιθανό, αρκεί οι κυβερνήσεις να κάνουν τα επισχυμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρέτσου, θέλετε και να πάρετε το λόγο. Ναι, δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, είμαι πεπισμένη ότι δεν πρόκειται για έναν διάλογο μεταξύ κοφών. Εδώ έχουμε έρθει για να ακούσουμε πραγματικά τις απόψεις σας, τις ανησυχίες σας. Ήρθα εδώ με τον συνάδελφό μου αντιπρόεδρο Κατάινεν ακριβώς για αυτό το λόγο για να ακούσω τους δικού σα προβληματισμού. Αλλά όχι για να πάρουμε αποφάσεις. Δεν γίνεται να λάβουμε αποφάσεις εξ ονόματο του Σώματος των Επιτρόπων, ούτε μπορούμε να πούμε ποια προγράμματα θα ανασταλούν, ούτε ποιο θα είναι το ποσό. Οι αποφάσει αυτές θα ληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού πρώτα συζητηθούν από το Σώμα των Επιτρόπων. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να λάβουμε τις ε, εκθέσεις των δύο χωρών οι δύο χώρε έχουν υποσχεθεί, έχουν δεσμευθεί να υποβάλουν σχέδια προπολογισμού ω τι 15 Οκτωβρίου. Γνωρίζετε κι εσείς ότι ε, βάσει με την εξαπλή δέσμη μέτρων, το SIXPAC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να έχει ζητήσει κύρωση 0,2% του ΑΕΠ. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν υποβάλει αίτηση ακύρωσης του προστίμου. Αυτό το πρόστιμο θα είχε πλήξει σοβαρά και μακροπρόθεσμα αυτές τις δύο χώρες. Στην επιστολή τους η Πορτογαλία και η Ισπανία επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους έως τις 15 ε, Οκτωβρίου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Καλό τον κύριο Ποστινάρου να μπει λίγο στη θέση μου, αν θέλετε. Εσείς, στη θέση μου, τι θα κάνατε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος υπέρμαχος ε, της περιφερειακής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής από μένα ιδίω σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ξέρω ότι στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη η πολιτική συνοχής έχει σχεδιαστεί ακριβώς με αυτό το σκοπό εξομάλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων. Και είναι ένα από τα βασικά μας και συνεχή μελήματα. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο εσείς εκπροσωπείτε τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών και όπως είπε ο κ. Κοτσολίνο, όλα αυτά είναι απόρρια της ε, νομοθεσίας που έχει υιοθετηθεί από, τους, ε, την προηγούμενη θητεία, από τους δύο συνομοθέτες. Μπορείτε να αλλάξετε τον κανονισμό, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Ο κ. Κοτσολίνο προέρχεται από μία περιφέρεια όπου η μακροοικονομική αιρεσιμότητα δεν εφαρμόζεται από την Νότια Ιταλία. Και με τα αναφέρω ότι εάν δεν τηρούνται οι αρχές της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, δεν θα υπάρξει και ανάπτυξη αυτής της περιφέρειας. Ξέρετε ότι υπάρχουν περιφέρειες όπου διοχετεύονται εκατομμύρια ευρώ όμως τελικά δεν υπάρχουν ε, απτές, ε, απτά ωφέλη στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Και υπάρχει μια ε, διασύνδεση μεταξύ του υπερβολικού ελλείμματος και της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Η αιρεσιμότητα λοιπόν έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να υπάρχει μια στρατηγική σε κάθε μία τέτοια περιφέρεια. Γιατί με, αυτές, με αυτή τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα μπορούμε να διαμορφώσουμε και μια στρατηγική για όλε τι χώρε για το ψηφιακό θεματολόγιο, τι επενδύσει σε όλου του τομεί. Επομένω, από πρακτική άποψη, όπω είπε ο κ. Γκουαλτιέρη, εγώ, σε αντίθεση μάλλον με αυτό που είπατε, κ. Γκουαλτιέρη, εγώ θεωρώ ότι είναι μια θετική πρόκληση αυτή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα για πολλέ αυτέ τι χώρε. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Δεν νομίζω ότι η Ιταλία θα είχε αναπτυχθεί και θα είχε ε, καταρτήσει πολιτική για τα ευρωζωνικά δίκτυα αν δεν είχαμε αυτή την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και υπάρχουν πολλά ακόμα παραδείγματα. Πολωνία. Στην Πολωνία λοιπόν υπάρχουν ε, θετικά κίνητρα για να διαμορφωθεί το πλαίσιο επενδύσεων και μεγιστοποίηση του αντικτύπου από αυτές τις ε, επενδύσεις ε, στις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους Επιτρόπους, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι. Αυτός ήταν ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων και συνομιλιών για το θέμα αυτό. Ήταν το πρώτο επίπεδο αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου και οι Επίτροποι άκουσαν πολύ σαφώς ε, το μήνυμα των μελών ε, τη Επιτροπής Ρέτζη. Και θέλω να τονίσω, εμείς τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη καταλαβαίνουμε το ρόλο μας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και το ρόλο μας για τη διατήρηση τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και την καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση. Καταλαβαίνουμε τη σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Θέλουμε όμως να μάθουμε τα πραγματικά στοιχεία, να γνωρίσουμε ποιες είναι οι συνθήκες ε, και να έχουμε την αναλυτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πώς ε, σκοπεύετε να ενεργήσετε στο μέλλον. Αυτό είναι το μήνυμά μας προς εσάς. Δίνω το λόγο στον συναδελφό μου, τον κύριο Γκουαλτιέρη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε λοιπόν τώρα στην ΕΚΟΝ. Τέσσερα λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για διάλογο, οπότε οι ευρωβουλευτές ε, θα ε, έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν κάποια δήλωση αν θέλουν, ε, να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε αυτήν παρά στην ερώτηση τους. Έχετε λοιπόν την ελευθερία να χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε το χρόνο σας. Ο Μπούρθαρ Πάλς είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο Κατάινιν ε, και την ε, ε, Επίτροπο Κρετή. Η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να υποβάλει πρόταση σχετικά με την αναστολή των ταμείων. Ε, όταν ε, τα κράτη δεν έχουν ε, καταβάλει καμία προσπάθεια για μείωση του υπερβολικού ελλείμματος. Και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τη διαδικασία της συναπόφασης έχουν υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία. Εμένα και άλλους προλαλήσαντες μας ενόχλησε το ότι υπόθηκε ως επιχείρημα ότι είμαι κατά επειδή πάντα ήμουν κατά. Εάν εμείς ως Κοινοβούλιο αρχίσουμε να λέμε ότι κάποτε στο παρελθόν ήμουν κατά κάποιου θέματος, ε, γι' αυτό δεν το θέλω και σήμερα, τότε θα ήταν πολύ δύσκολη η συνεργασία μας εδώ. Και οι συνάδελφοι εδώ μπροστά νομίζω το διατύπωσαν πολύ σαφώς. Πρόκειται λοιπόν για εξουσιοδότηση όχι για τρέχοντα προγράμματα, όπως είπε πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μιλάμε για μελλοντικά προγράμματα. Και κατά τη γνώμη μου, δεν μιλάμε για ακύρωση των ταμείων, αλλά για πιθανή και τονίζω πιθανή αναβολή, αναστολή. Δηλαδή, τα ταμεία για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση αναστολής μπορεί αργότερα να απελευθερωθούν. Η σχετικοί πόρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομίζω επαρκείς δυνατότητες να εξετάσουν το πώς, πότε ε, και ε, το πώς και το πότε της αναστολής. Και θα ήθελα λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει σαφώς διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ισπανία βρίσκεται σε, σε κάποιον δρόμο, ενώ δυστυχώς δεν βλέπω τέτοια κατεύθυνση από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, την νέα κυβέρνηση. Οι συνθήκες πλαίσιο για την αναστολή των πληρωμών ε, θα πρέπει να αποφασιστεί με αντικειμενικά κριτήρια. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι δίκαιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση. Επαναλαμβάνω όμως ότι βασίζομαι στη σοφία της Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να υποβάλει τέτοια πρόταση. Εγώ προσωπικά, και θα ήθελα να το πω αυτό σαφώς, διότι αυτή είναι η θέση μου και πολλών άλλων στην, στην πολιτική μου ομάδα, δεν θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παραβεί τους κανόνες. Ε, βλέπω ότι ε, μου μένει λεπτό ακόμα να δώσω την ευκαιρία λοιπόν στην Κομισιόν να απαντήσει. Θα με ενδιαφέρει επίσης πότε σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τέτοια πρόταση. like to... Ποιος θα ήθελε να απαντήσει. Πολύ σύντομα. Για την τελευταία ερώτηση, πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη, δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα. Έτσι λοιπόν, ε, μαζί με την ε, συνάδελφο Κρέτσου θα κάνουμε μια αναφορά αύριο στους συναδέλφους στην Κομισιόν και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Όμως, ε, σωστά είπατε ότι αν υπάρχει μια Αμερική αναστολή μπορεί και θα, πρέπει να έρθει αμέσως αφού θα έχει αναλύσει η Κομισιόν ότι ακολουθεί τη δημοσιονομική οδό η χώρα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα πρέπει, θα πρέπει να γίνει άμεση άρση. Κύριε Μπάλτς, ο κύριος Μπάλτς είπε ε, κάτι διαφορετικό, γιατί μίλησε και για το πότε ε, όταν θα γίνει η πρόταση, γιατί αν έχω καταλάβει καλά δεν υπάρχει προθεσμία στον κανονισμό για το πότε υποβάλλουμε την πρόταση, δεν είναι πουθενά γραμμένο. Και η Επίτροπος Κρέτσου είπε ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο μετά την απόφαση στην παράγραφο 10. Αλλά δεν λέγεται ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία πουθενά στον κανονισμό. Κυρία Περβανσπρές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι εδώ φαίνεται πόσο σημαντικό είναι αυτός ο διαρθρωτικός διάλογος. Αγωνίστηκε πολύ το Κοινοβούλιο για να τον εντάξει στην νομοθεσία, γιατί νομίζω ότι αποδεικνύουμε εδώ σε μια οικονομικοπολιτική και νομική και λογιστική συζήτηση για την πράγμα μιλάμε. Κύριε Κατάινεν, γιατί ο κύριος ε, την και εσείς που είστε μας ε, απόψε, ε, και ταυτόχρονα στη Λισαβόνα ανακοίνωσε ότι χρειάζεται η Πορτογαλία ένα νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής βοήθειας, κοινωνικονομικής βοήθειας, ε, γιατί πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Είστε αρμόδιος επίτροπος κύριε Κατάινεν για τις επενδύσεις κατά κάποιο τρόπο και αν δούμε την κατάσταση στις δύο χώρες και δύο στην Πορτογαλία βλέπουμε ότι στην Πορτογαλία ε, υπάρχει ουσιαστικά μια ανάγκη να απαντήσουν στις απαιτήσει του Συμφώνου Σταθερότητας και του ΣΥΚΣΠΑ και αυτό θέτει σε μια ευάλωτη κατάσταση της επενδύσεις. Ε, τώρα πρέπει να δούμε λοιπόν αυτή την ευρωπαϊκή ικανότητα επενδύσεων, ιδίω μέσα των διαθροτικών ταμείων, γιατί όπως ξέρετε, λαμβάνοντα υπόψη το επίπεδο του δημόσιου και του ιδιωτικού κρέους, στην Πορτογαλία είναι πολύ μικρά τα περιθώρια για τις επενδύσεις και αν ε, δούμε και ε, το σχέδιο ΕΦΣΥ ε, στο οποίο από κοινού έχετε εκπονήσει με τον κύριο Γιούνκερ, αυτό ε, δεν μπορεί ε, ουσιαστικά να τροφοδοτήσει ιδιαίτερα την πορτογαλική οικονομία, γιατί από τα 10 δις έχει πάρει ένα πολύ μικρό ποσό η Πορτογαλία. Και είπατε, και το είπε και η κυρία Κρέτσου, ε, είπατε ότι δεν είναι τόσο σοβαρό γιατί θα ήταν προσωρινά τα μέτρα ε, και δεν θα έχουν ε, βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο. Όμω όταν μιλάμε για μια τόσο εύθραστη, μια τόσο ευάλωτη οικονομία η οποία επίση κινητοποιείται για να ανακάμψει οποιοδήποτε αρνητικό μήνυμα δοθεί στους επενδυτές υποσκάπτει αυτό το τόσο απαραίτητο κλίμα που χρειαζόμαστε να είναι φιλικό για τις επενδύσεις. Και ας δούμε την κατάσταση της Πορτογαλίας. Ε, θα έχει ένα έλλειμμα 2,5% Πορτογαλία. Τι παραπάνω θέλετε. Επί της δεν έχετε πάρει την απόφασή σας ε, και χαιρόμαστε ε, για το ότι υλοποιούμε αυτό τον διαρθρωμένο διάλογο εδώ. Θα μπορούσα ίσως να σας προτείνω το εξής γιατί θα πρέπει φυσικά να σεβόμαστε και τους κανόνες και να αναλύουμε και τον παραλληλισμό των τύπων. Καθώς το Συμβούλιο εκτίμησε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μηδέν κυρώσεις, ε, ε, θα μπορούσατε να ακολουθήσετε και τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου που σας προτείνει και μηδενική αναστολή γιατί ακούω κι άλλο ένα επιχείρημα που λέει «Α, θα προβούμε σε αναστολή και μετά ε, στο 2017 θα έχουμε θετικές δράσεις και θα σταματήσουμε την αναστολή». Για την αξιοπιστία της Κομισιόν, ειλικρινά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τον προπολογισμό που θα σας παρουσιάσουν και να δείτε αν πρέπει να προχωρήσετε στην αναστολή. Αν ε, πράγματι δεν θέλετε τώρα εδώ απλό να ακολουθείτε ε, τους ε, τύπους έχετε ουσιαστικά ε, αυτές τις λύσεις που τις διερευνάτε αυτή τη στιγμή και ελπίζω να μπορέσετε να λάβετε υπόψη την νομοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωραία. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, αλλά σίγουρα θα υπάρξει χρόνος ε, απαντήσεων. Ε, ο Μπεντλούκα για το ECR. Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στην, στην ε, δήλωση της Κομισιόν ότι μιλάμε εδώ για αναστολή των ε, υποχρεώσεων ε, και όχι των πληρωμών. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά αφελές, διότι φυσικά θα ε, καθυστερήσουν επενδύσεις, θα αυξηθεί ο κίνδυνος για τους επενδυτές εάν γνωρίζουν ότι η συγχρηματοδότηση εξαρτάται από το κατά πόσο η κυβέρνηση της χώρας τους πληρεί τις υποχρεώσεις τους και ε, βλέπουμε ότι συχνά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η αναστολή αυτή λοιπόν φυσικά θα οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων. και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθούν εδώ, ότι το ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα είναι λάθος. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να περιορίσουμε την κατανάλωση και όχι τις επενδύσεις σε, σε ε, μειονεκτικές περιοχές. Και Εάν αναφερθεί κανείς στον ευρωσκεπτικισμό, νομίζω ότι θα αυξηθεί ο ευρωσκεπτικισμός εάν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραβεί τους κανόνες ε, του. Και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους κανόνες. Εάν ανασταλούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, τότε ε, τι γίνεται με την ε, περιφερειακή πολιτική. Φυσικά μπορούν τα κράτη-μέλη τους πόρους από την κατανάλωση να τους μεταφέρουν ε, σε επενδύσεις. Και προσωρινά, όπως πιστεύει ο κύριος Κατάινεν, ή μόνιμα να αντικαταστήσουν τους πόρους αυτούς. Ε, και έτσι νομίζω ότι έχουμε καλύτερο τρόπο δαπάνης των χρημάτων και για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η δυνατότητα να προβλέψει την καλύτερη δυνατή κατανάλωση των ε, πόρων, δαπάνη των πόρων, αυξάνοντας τη το ποσοστό συγχρηματοδότησης που πρέπει να δίδεται από τρίτους ώστε να μπορέσουν να μειωθούν μέρη του Ταμείου Συνοχής, αλλά για κάθε πρόγραμμα να παραμένει ένα ποσοστό χρηματοδότησης από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα οδηγούσε ε, στη χρηματοδότηση προς ε, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα, διότι ε, έχουν επιδείξει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Όταν Βλέπω τι γίνεται στην Ελλάδα με το 100% της χρηματοδότησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, χωρίς ε, δηλαδή συγχρηματοδότηση. Μήπως θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό συγχρηματοδότησης από τρίτους. Η ε, ερώτησή μου είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σκέφτεται αυτό, διότι νομίζω ότι θα χρειαστεί ε, καθοδήγηση όσον αφορά τη δαπάνη των περιφερειακών πόρων. Ευχαριστώ. Θα θέλατε να σχολιάσετε, κύριε Κατάινεν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, σίγουρα δεν θέλω να σχολιάσω. Ε, τα όσα έχουν, ακουστεί για το μέλλον της, Πολων... της ε, Πορτογαλίας. Δεν θέλω καθόλου να το σχολιάσω αυτό. Κοινή μας πρόθεση είναι να στηρίξουμε την Πορτογαλία για να προοδεύσει και να έχει βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν ε, χρειάζονται αυτή τη στιγμή μηνύματα αποσταθεροποίησης. Δεύτερη παρατήρηση. Η κυρία Περές είπε ότι η Πορτογαλία χρειάζεται κάθε δυνατό μέσο για υποστήριξη των ε, δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Συμφωνώ πολύ με αυτό. Δεν θέλω να προδικάσω τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν όμως αποφασίσουμε να δαπανίσουμε μέρος ε, των αναλήψεων υποχρεώσεων, ε, θα υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση προς τη χώρα. Επίσης, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ε, μη απορροφημένων υποχρεώσεων και θα υπάρχουν ακόμα σε περίπτωση μερικής αναστολής. Η χώρα δεν έχει καταφέρει να απορροφήσει πολλούς πόρους ε, κατά τη διάρκεια αυτής της προγραμματικής περίοδου. Όσον αφορά την μηδενική αναστολή και την πρότασή σας, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορώ να προδικάσω καμία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή. Μία τελική παρατήρηση. Όσον αφορά την ε, χρονική προοπτική, η Πορτογαλία και η Ισπανία θα υποβάλουν ε, σχέδιο προϋπολογισμού στις 15 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τα προγράμματα αυτά, όπως, τους προϋπολογισμούς αυτούς, ε, όπως αξιολογεί τον προϋπολογισμό κάθε χώρας. Και ας υποθέσουμε ότι υπάρξει απόφαση μερικής αναστολής. Μόλις διαπιστώσουμε ότι οι χώρες αυτές ε, πληρούν τις υποχρεώσεις τους, ε, τότε θα μπορέσουμε να άρουμε την αναστολή. Αυτή είναι η λογική. Η απόφαση για ε, αναστολή μπορεί να ληφθεί ε, τώρα το φθινόπωρο, και, αλλά και η απόφαση για άρση μπορεί να ληφθεί επίσης μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο. Η Σιλβί Κουλάρ. Είναι αδικό. Είχα αφήσει κάποιο χρόνο για να απαντήσει ο Επίτροπος στην ερώτησή και χρησιμοποιείται ε, και τώρα ο χρόνος για να απαντηθεί η ερώτηση των άλλων ομιλητών. Αν έχουμε κανόνε, θα πρέπει να του στηρίσουμε. Θα πρέπει η Κομισιόν να απαντήσει σε ερωτήσει Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να περάσουμε στην κυρία Σιλβιγκουλάρ. Συμφωνώ όμω ε, ότι ο κάθε ε, Ευρωβουλευτή θα πρέπει να λάβει και την απάντησή του. Ε, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, είναι πολύ καλή ε, και σα Σας, ευχαριστώ, συμβολίζει με ιδιαίτερο τρόπο την κατάσταση του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να επιλέξουμε το στρατόπεδό μα. Δεν είναι ότι έχουμε κανόνε που υπάρχουν και δεν θα πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να διαλέξουμε μεριά. Με αυτού που θέλουν αυστηρού ή ευέλικτου κανόνε. Είμαστε στη δεξιά ή στην αριστερά. Αλλά έτσι θα πάμε και πολύ μακριά. Ε, θα θέσω τρία-τέσσερα σημεία προβληματισμού στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουμε, θεωρώ. Πρώτον, ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε εδώ ότι ο αντίκτυπος ε, της κρίσης ε, στις εν λόγω χώρες ε, χρήζει εξέτασης σε ανθρώπινο επίπεδο. Από κοινού δημιουργήσαμε την Ευρώπη, όχι για να τιμωρήσουμε τους πολίτες που μάλιστα πλήττονται από την κρίση και ξεχνάμε κάποιες φορές ότι υπάρχει και περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επομένως, όλους μας αφορά η, τα βάσανα του καθελαού η ανέχεια, η ανεργία ε, σε όλες τις χώρες. Μετά, πρέπει να έχουμε κατά νου και την ε, έλλειψη αξιοπιστία σε όλη την Ευρώπη, από το βορρά μέχρι τον νότο, γιατί υπάρχουν και χώρες που... Ε, συμβάλλουν, υπάρχουν Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που θα πρέπει να έχουν την εντύπωση ότι πολύ σωστά δαπανώνται τα χρήματά τους. Και θεωρώ αρκετά κομικό μάλλον να λέμε και στερεοτυπικό να λέμε ότι υπάρχουν ε, πλούσιοι στο βορρά και φτωχοί στο νότο. Παντού υπάρχουν φορολογούμενοι που συμβάλλουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τρίτον, η σημασία των κανόνων. Είναι κάτι εκπληκτικό. Λε και δεν ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτοί οι κανόνε. Λε και δεν εξετάσαμε. Για να δω. 450 τόσοι ψήφοι υπέρ. Και έχουμε και τον ε, εισηγητή ε, σε ό,τι αφορά το six-pack. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να είναι ε, πιο αντικειμενική και να μην κάνει καμία εξαίρεση. Επομένω, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τι θα πάρει ο καθένα από την Ευρώπη, αλλά και τι μπορούμε να συμβάλλουμε στην Ευρώπη. Προσπαθεί να βρει τρίτο δρόμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ σα ενθαρρύνω να προσπαθήσετε σε αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρημα γιατί πρέπει, εγώ σας καλώ να ε, τηρήσετε τους κανόνες αλλά και να τους εφαρμόσετε με έξυπνο τρόπο για να έχει ώστε το μικρότερες επιπτώσεις για το μέλλον. Ποια θα είναι λοιπόν η επίπτωση για το μέλλον. Κάποιοι λένε ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις για τα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει ήδη. Όμως, με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται, γίνεται να προβλέψουμε να έχει το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο μέλλον. Γιατί οι επενδύσεις πάντα είναι στραμμένες προς το μέλλον και εμείς θέλουμε η Ευρώπη να έχει ένα μέλλον. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να διευκρινίσω, όπως είπε και ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπουν ε, τα ευρωπαϊκά ταμεία, δεν υπάρχει καμία προθεσμία για την αναστολή των κονδυλίων αυτό από την άλλη. Είμαι πεπισμένη όπως και εμείς και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένουμε φυσικά και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μια σύσταση, όπως είπε η κυρία Πέρες. Και όπως σας είπα, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη τις δικές σας προτάσεις ε, και ίσως και θα αποφασίσουμε μετά από τα προσχέδια προπολογισμού που θα υποβάλουν οι δύο χώρε Όμως φυσικά δεν εξαρτάται από του τους δύο να αποφασίσουμε. Θα είναι μια απόφαση που θα ληφθεί από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μου άρεσε η ιδέα σας ε, περί ανθρώπινης προοπτικής. Ε, δεν κάνουμε πολιτική, Κάνουμε πολιτική για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και η πολιτική της συνοχής νομίζω ότι είναι η πιο απτή πολιτική και ορατή πολιτική που δείχνει πώς μειώνονται οι ανισότητες. Και χαίρομαι πάρα πολύ για όσα είπατε για τις ε, διαφορές και το χάσμα μεταξύ Ανατολής, Δύσης, Βορρά, Νότου. Νομίζω είναι επικίνδυνη αυτή η οδός. Είναι λοιπόν προφανές ότι η λιλεγγύη θα πρέπει να συνάδει με την ευθύνη. Έχουμε νομοθεσία και θα πρέπει να την εφαρμόσουμε. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, οι χώρες αυτές είχαν ε, πολύ μεγάλα ποσά που δεν είχαν δαπανίσει από το 2014, το 2015 και το 2016 από τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων αυτών των ετών. Αν υπάρχει λοιπόν αναστολή, θα είναι ένα μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2017 και δεν αναμένω. Είμαι σίγουρη ότι οι δύο αυτές χώρες ε, δεν θα περιμένουν μέχρι το 2020 ε, όταν ε, θα εμφανίσουν τα αποτελέσματα αυτής της αναστολής. Έτσι λοιπόν σας διαβεβαιώ ότι δεν θα χαθεί ούτε σέντ. Όμως είναι αυτή η ευαισθησία ένα πολιτικό μήνυμα και φυσικά έχει και συμβολική αξία. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητας να σεβαστούμε τους κανόνες που υιοθετούνται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και φυσικά της εικόνας που δίνουμε στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, εγώ ειλικρινά θεωρώ ότι αρχίσαμε αυτό το διάλογο και ακούω την θέση που εκφράστηκε στην αρχή. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει μια τεράστια φάρσα αυτή εδώ. Ε, καθώς ε, δεν ε, εκλέγεται η Επιτροπή από τους πολίτες, ε, τελικά θα λάβει μια απόφαση που θα αποτελέσει έγκλημα έναντι ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ξέρετε ότι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι ε, υπέφεραν ε, τις συνέπειες για πολλά χρόνια μίας ε, ηλίθιας λιτότητας και ακόμη πληρώνουν τις συνέπειες. Ο κύριος Κατάνινεν μίλησε εδώ για την αστολή των κονδυλίων σαν να ήταν κίνητρο. Δεν είναι κίνητρο. Ξέρω ότι μιλά μια περίεργη γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν είναι κίνητρο αυτό σε πολλούς από εμάς δεν μας αρέσει η δουλειά που κάνετε εσείς ή ε, οι συναδελφοί σας. Αν ε, εμείς ε, αναστέλαμε ως κίνητρο το μισό μισθό σας, θα το θεωρούσατε ότι είναι κίνητρο ή κύρωση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το κίνητρο στην γλώσσα της Κομισιόν. Αυτό που κάνετε είναι ότι μας αντιμετωπίζετε με κινησμό. Ε, και ουσιαστικά μια τιμωρία παρουσιάζει το κίνητρο, αλλά δεν είναι. Αυτό που προτείνεται εδώ από την Κομισιόν σήμερα στις δύο χώρες, που ήταν οι δύο χώρες που τιμωρήθηκαν περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που τους προτείνεται ε, είναι να τιμωρηθούν, να του επιβληθούν παράλογες και αντιπαραγωγικές κυρώσει που είναι εντελώ άδικες και αφού υποχρεώθηκαν να μειώσουν τα ποσοστά επενδύσεων και σχεδόν τίποτα γιατί όλες οι επενδύσεις έφτασαν ε, το ελάχιστο ρεκόρ και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία εσείς θέλετε τώρα να παρουσιάσετε αντιπαραγωγικές ε, κυρώσεις έτσι λοιπόν αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και δεν έχει σημασία πόσο θέλετε να χρυσώσετε το χάπι. Έτσι λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο στόχο. Εδώ προετοιμάζεται μια μόνιμη διαδικασία σαμποτάζ. Θέλετε να διατηρήσετε αυτέ τι χώρε σε μια μόνιμη ευάλωτη κατάσταση για να μπορεί η Κομισιόν να επιβάλλει κάποιε επιλογέ που ο λαό απέρριψε, ιδίω στην Πορτογαλία. Έτσι λοιπόν, αυτό θέλετε να κάνετε με αυτούς τους λαούς να πρέπει να δεκτούν κατάχρηση και δεν, να τους ε, επιτρέψετε να σηκώσουν το κεφάλι και να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε ελπίδα ε, μπορεί να υπήρχε στο ευρωπαϊκό οικονομήμα και είναι συνώνυμη της ε, αλληλεγγύης καταστρέφεται τη στιγμή που θα αποφασίσει η Κομισιόν την αναστολή των διαφορετικών ταμείων. Αν ψηφίσετε ουσιαστικά θα μας δείξετε τη μετριότητα της ευρωπαϊκής ε, ηγεσίας. Ξέρω ότι ε, εσείς ε, θα γραφτείτε στην ιστορία ως ε, άνθρωποι που έχουν, επιζη... που έχουν δράσει επιζήμια για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Ευχαριστώ. Βέβαια, επιμένω να αφήνετε και χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. στο το για τους πρασίνους. Καλησπέρα. Είναι προφανές ε, το αίσθημα που κυριαρχεί εδώ ότι δεν θα πρέπει να ελοπιθεί κάτι τέτοιο. Ε, εγώ θα ήθελα να πω λίγο πιο πίσω, κύριε Επιτροπή, στο πώς κυλήσει η συζήτηση στις διαπραγματευτικές ε, ε, στις διαπραγματεύσεις της δημοσιονομικής με την Ισπανία. Εσείς ε, ουσιαστικά είχατε ε, παρακολουθήσει την όλη διαδικασία γιατί στο διάλογο που είχαμε μαζί σας σας είχαμε επισημάνει ότι η δημοσιονομική μεταρρύθμιση ε, στην Ισπανία θα παρεκκλίνει και ότι δεν θα πετύχει η εργασική μεταρρύθμιση. Είχατε στρέψει το βλέμμα σας αλλού επειδή ήταν εκλογική χρονιά κτλ. Όμως η ανεξάρτητη φορολογική αρχή τα έλεγε στη Μαδρίτη ότι δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα και είχαμε φέτος μείωση των φορολογικών εσόδων από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο της τάξης του 8% και τελικά συσκητούσατε από την άλλη πλευρά και ε, τελικά τι κάνετε, κοιτάτε από την, μία, από άλλη πλευρά σε μία περίπτωση και έρχεστε να τιμωρήσετε αυτούς που δεν φταίνε, έρχεστε να τιμωρήσετε τους πολίτες που δεν φταίνε τίποτα και τελικά τι κάνετε, αυτό κάνετε και δίνετε κίνητρα σε όποιον δεν σέβεται τα συμφωνηθέντα. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά μία καυκιακή κατάσταση. Ε, πρέπει ουσιαστικά να σκεφτούμε ε, τι ακριβώς κάνουμε με τα μέτρα φαίνεται σαν να εφαρμόζονται τα μέτρα, αλλά καθώς ε, δεν γίνεται να εφαρμοστούν, δεν θα τα τηρήσω. Ε, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να αρχίσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και θα ήταν καλό να επισημάνουμε ότι εσείς ε, ε, με τη δική σας διακριτική ευχέρεια εφαρμόζετε τα μέτρα. Γιατί η Κομισιόν, παραδείγματος χάρη, πάντοτε επιβάλλει κυρώσεις βάσει του ελίμετος και δεν το κάνει βάσει της διαδικασίας της μακροοικονομικής διαδικασίας ανισορροπιών και θέλω να επισημάνω και τρία πράγματα. Καταρχήν, θέλω να σας ρωτήσω αν θα κάνετε μία μελέτη για τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η αναστολή κάποιων κονδυλίων. Δεύτερον, υπάρχει κάτι που με εξέπληξε, είπατε κυρία Κατάινεν, ότι δεν συμβαίνει τίποτα γιατί περσεύουν τόσα πολλά χρήματα, έχουν απορροφήσει τα κράτη τόσο λίγα κονδύλια και ακόμη και αν υπάρχουν κυρώσει θα εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Εσεί έχετε προγράμματα για να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη να απορροφούν τα κονδύλια ε, και αναγνωρίζετε ότι είναι εντελώ αποτυχημένα αυτά τα προγράμματα ή δεν τα εμπιστεύετε. Και αν μα λέτε κάτι τέτοιο, τελικά σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεστε τα προγράμματά σα. Ένα λεπτό σα έχει μείνει. Ναι, ναι, το ξέρω. Βλέπω το χρόνο, Ρομπέρτο. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν, πιστεύετε σε αυτά τα προγράμματα και αν δεν απαντήσει εντάξει, είναι μια δήλωση απλώς. Και μπορώ να έχω τις απαντήσεις αργότερα και κάτι τελευταίο. Αυτό για τους συναδέλφους που έχει για σας. Όλοι συμφωνούμε στο ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα ε, ουσιαστικά ε, είναι αρνητική και γιατί δεν κάνουμε ένα ψήφισμα και να ζητήσουμε μπλοκάρισμα από το Συμβούλιο εδώ. Ε, η Κομισιόν έχει την νομική υποχρέωση να πυροδοτήσει τη διακασία, όμως το Συμβούλιο μπορεί να τον μπλοκάρει και ζητώ εγώ λοιπόν να ζητήσουμε από το Συμβούλιο κάτι τέτοιο. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Κατάινεν. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να απαντήσω σωστά στις ερωτήσεις σας μέσα σε 11 δευτερόλεπτα. Έχουμε βελτιώσει την τεχνική μας βοήθεια για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να απορροφήσουν ε, τα τους πόρους των διαφορετικών ταμείων. Ε, και μάλιστα έχουμε φτάσει σε τελείως διαφορετικά επίπεδα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Όπως είπα νωρίτερα, Κανείς δεν θα χάσει ούτε, ούτε ούτε λεπτό, εάν ε, οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αυτά που πρέπει και πρέπει να τα κάνουν αυτά όχι επειδή το επιβάλλει η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή θα βοηθήσουν τι χώρε ε, να ξαναβρεθούν στον χώρο τη ανάπτυξη. Μόνο κάποιο που πιστεύει ότι ε, οι δύο χώρε αυτέ δεν θα κάνουν όσα έχουν υποσχεθεί στου πολίτε του ε, θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, Μαρκο από το EFTD. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι ούτε Πορτογάλο ούτε Ισπανό, είμαι Ιταλό και ανήκω σε αυτές τις χώρες ε, που έχουν προσυπογράψει δυστυχώς ε, αυτούς ε, τους κανόνες και δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία που δεν σέβονται τους κανόνες και τι κάνει η Κομισιόν ουσιαστικά μπλέκει όλη την οικονομία των χωρών της Νότιας Ευρώπης και πάει και επιβάλλει εδώ ε, συζητούμε ε, για κάποια λεπτομερία ενώ έχουμε πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα που συνδέεται με την ΟΝΕ και δεν το λύνουμε και τελικά οι κανόνες μεγεθύνουν αυτό το πρόβλημα καθώς επιβάλλουν λανθασμένες κυρώσεις, δηλαδή επιβάλλουν τις ε, κυρώσεις της χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας και αντίθετα οι χώρες που προκαλούν ανισορροπίες όπως ε, οι κάτω χώρες η Γερμανία στο ισοζύγιο πληρωμών αυτές ε, έχουν διαδικασίες που τις ευνοούν περισσότερο, όπως και η Γαλλία. Έχουμε τα λόγια του Γιούν και η Γαλλία είναι η Γαλλία, κάνει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, όμω, ε, από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργούν οι κανόνε. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο οικονομικό και νομισματικό πρόβλημα. Ο Στίγκλιτς ε, ουσιαστικά έκανε μια προειδοποίηση φέτο το καλοκαίρι και είπε ότι αν ε, δεν δώσουμε προσοχή στη νομισματική ένωση και σε μια οικονομική περιφέρεια που δεν είναι ολοκληρωμένη και κάνουμε λανθασμένε μεταρρυθμίσει μισθολογικού τύπου, παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, θα επιζήσει πέρα από τη σημερινή θητεία. Έτσι λοιπόν εδώ είναι το θέμα. Μια νομισματική πολιτική δεν μπορεί να πηγαίνει καλά για 19 χώρε που έχουν διαφορετικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Θα πρέπει να σταματήσουμε να υπερασπίζουμε την ορθοδοξία αυτού του εργαλείου και να αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά πριν να φτάσουμε σε ανεξέλεκτη κατάσταση ε, γιατί ε, η Ευρώπη θα πρέπει να διαχειριστεί κάτι τεράστιο που θα είναι και ανεξέλεγκτο. Έτσι λοιπόν, εγώ προτιμώ να κάτσω στο τραπέζι και να πω που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προς την ε, ΟΝΕ, να κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω, αλλά εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε σε ηλίθιες κυρώσεις και που σε κάποιε χώρε που είναι ισχυρέ δεν εφαρμόζεται, γιατί αυτό γίνεται. Έχουμε τα χρήματα ιδρύματα ε, της Γερμανίας που καταλήγουν να χρηματοδοτούν τις διάφορες μελέτες κτλ. Και κανείς δεν κάνει τίποτα. Ενώ όταν πρόκειται για φτωχέ και αδύνατες χώρες, εδώ είστε ισχυροί εσείς της Κομισιόν. Αυτό αντιλαμβάνονται οι πολίτες αυτή τη στιγμή. Πολύ σύντομα όλοι συμφωνούν ότι οι άνθρωποι στην Ισπανία και την Πορτογαλία έχουν υποφέρει πολύ τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τραγωδία για τους απλούς ανθρώπους που έχασαν τις δουλειές τους και την ελπίδα τους για το μέλλον. Είδαμε όμως και κάποια ενθαρρυντικά σημάδια. Για παράδειγμα, η ισπανική οικονομία αναπτύσσεται πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα ε, αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται όμως παρόλα αυτά περισσότερες θέσεις εργασίας ε, και χρειαζόμαστε σταθερότητα. Και η σταθερότητα θα επέλθει όταν ε, θεωρήσουν οι άνθρωποι ότι η χώρα έχει ξεφύγει από τα προβλήματα. Επίσης, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη βασίζεται στο κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε ως, ε, με, βασική αρχή το κράτος του δικαίου, κάτι που αντικατέστησε την εξουσία του πιο ισχυρού. Το κράτος δικαίου βασίζεται στο καθένα να εκπληρεί τι υποχρεώσει του. Είμαστε αλληλέγγυοι, θέλουμε να βοηθήσουμε και ο καθένα πρέπει να φέρει το βάρο του. Εάν δεν εμπιστευόμαστε ο ένα στον άλλον, δεν μπορεί να υπάρξει αλληλεγγύη και δεν μπορεί να υπάρξει ένωση ιδανικών. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθήκων θα πρέπει να φροντίσει να ε, εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ακόμα και αν υπάρχει πολιτική βούληση να ε, παραβιάσουμε τους κανόνες δεν θα το κάνουμε αυτό, διότι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ενότητα. Εάν κάποιο θέλει να αλλάξει τους κανόνες τότε ναι. Η υποχρέωσή μας όμως είναι να φροντίσουμε οι κανόνες να εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε, και πάλι ε, προσπαθούμε να δώσουμε την εντύπωση ότι υποκαθιστούμε τα κράτη-μέλη. Εσεί μιλάτε για διευθυντικά ταμεία, όμω κρύβεται η ίδια πραγματικότητα, μεγαλύτερη απορρίθμιση και δέσμευση του εθνικού πλούτου. Είναι αυτό ο φιλελευθερισμό ε, ε, του βρυξελιώτικου μοντέλου που επιβάλλεται από τη Γερμανία με ενιαίο νόμισμα και νέα πολιτική. Σήμερα, από την επίπεδο στράγο είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία. 28 δις είπατε για την Ισπανία, ακριβώ το ποσό του φακέλου που θέλετε ακριβώς να παγώσετε για το 2014-2020. Ε, ε, ακριβώς θέλετε λοιπόν να μπλοκάρετε ε, την μελλοντική ανάκαμψη της ισπανικής οικονομίας. Είναι ένας θεσμικός εκβιασμός των Βρυξελών. Πρόκειται για μια άρνηση των, του σκοπού ακριβώς των Διευθυντικών Ταμείων και μείων Συνοχής, όμως ε, βλέπουμε ότι έχουν αυτόνομη ε, λογική και αυτόνομους κανόνες. Τώρα εδώ ακολουθείται μια πολιτική ε, λιτότητα που μάλιστα είναι καταπιεστική. Τώρα για τη συγχρηματοδότηση πλέον θα είναι μη επιχειρησιακά όλα αυτά τα προγράμματα. Είναι παράλογο λοιπόν να ε, ζητάτε τέτοια πράγματα από αυτές τις χώρες. Μην κάνετε τίποτα λοιπόν που να αντιβαίνει στα κονδύλια της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στα τελευταία ταμεία. Αυτοδιάθεση λοιπόν να έχουν αυτές οι χώρες ε, την ε, κυρίαρχη θέση τους ε, με τα σύνορά τους, τον προπολογισμό τους, τα συστήματά τους και δεν χρειάζεται να μου δώσετε απάντηση. Αν μπορώ να σχολιάσω γι' αυτό το ζήτημα αξιότιμο μέλο. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει ε, ουσιαστικά ε, να καταστήσει αιρέσιμα τα διευθυντικά ταμεία βάσει της πολιτικής λιτότητας. Δεν υπάρχουν όμω περιθώρια λιγμών, γιατί τα διαθετικά ταμεία έχουν και εξάντε και εξπόστε ερεσιμότητα. Είπατε ότι έχουν τη δική του νομική βάση. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι σε αυτό, αρκεί να διαβάσετε τον κανονισμό όπως έχει διατυπωθεί. Η εξάντια ερεσιμότητα λοιπόν για να λειτουργήσουν σωστά τα διευθυντικά ταμεία. Εξπόστε ερεσιμότητα για να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη να βάλουν τάξη στα δημόσια οικονομικά του και έτσι να αξιοποιηθεί στο έπακρο, ε, στο έπακρο τα κονδύλια που δαπανώνται από τα λεφτά του φορολογουμένου. Είπατε επίση ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τη δική του πολιτική και να μην υπάρχει ε, καμία ε, τραπεζική επίβλεψη ή άλλο τέτοιο κοινό μηχανισμό. Όμω τότε δεν θα υπάρχει ευρωπαϊκή οικονομία, κατά τη γνώμη μου, γιατί βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, αλλά και ε, στην έκθεση που υπάρχει από τον ένα στην οικονομία του άλλου. Επομένω, ε, μια πυρκαγιά σε ένα κράτο μέλο θα περάσει τα σύνορα ενεργείου οφθαλμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρεις σκέψεις να εκφράσω. Καταρχάς, πιστεύω ότι είναι ανησυχητικό το ότι αρκετοί ευρωβουλευτές εδώ πιστεύουν ότι τα κράτη-μέλη δεν θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας ε, υπερβολικού ελλείμματος. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτό δεν είναι ευθύνη ούτε του Κοινοβουλίου ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι ευθύνη των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων στις χώρες αυτές. Και εμείς έχουμε περάσει δύσκολες ε, στιγμές, αλλά εάν επιλέξει κανείς ε, να μειώσει τη χρηματοδότηση σε δύσκολες εποχές, ε, τότε υπονομεύει τις επενδύσεις. Δεύτερη παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση νομοθεσίας. Όταν λοιπόν νομοθετούμε, νομίζω ότι μπορούμε να απαιτήσουμε από όλους μας να ακολουθήσουμε τους κανόνες αυτούς, αλλιώς δεν τους χρειαζόμαστε και δεν είμαστε ένωση. Έχουμε κανόνες σχετικά με το πώς πληρώνει κανείς το τέλος της συμμετοχής του και τα διαφορετικά πληρώνουν διαφορετικό ποσό. Έχουμε επίσης κανόνες περί δημοσιονομικής σταθερότητας. Έχουμε κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που δεν ακολουθούνται αυτοί οι κανόνες αυτοί και έχουμε κανόνες που διέπνονται διάφορα ταμεία. Εάν εμείς ως Κοινοβούλιο Υπονοούμε ότι νομοθετήσαμε, αλλά δεν το εννοούσαμε και πολύ σοβαρά. Επρόκειτο απλά για μια δήλωση. Τότε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπονομεύουμε την αξιοπιστία όχι μόνο του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι υπονομεύουμε στην πραγματικότητα την ευρωπαϊκή οικονομία. Διότι αν ε, δεχτούμε ότι τα προβλήματα σε ένα κράτος μέλος θα λυθούν ε, με, αν έχουμε όλο και μεγαλύτερο έλλειμμα, τότε ε, θα έχουμε ανεργία και έλλειψη επενδύσεων. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε ή μάλλον κύριοι Πρόεδροι, το ερώτημα είναι Εάν το ερώτημα είναι αν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να στηρίζει το κράτο δικαίου, τότε υπάρχει μόνο μία απάντηση. Μπορούμε να συζητήσουμε τι θα γίνει με τι αναστολέ, αλλά θα πρέπει επίση να έχουμε κατά νου ότι υπολογίζουμε οι αλληματικέ χώρες να πληρούν τις, διαδικασίες τους, τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας. Και αν κάποιοι εδώ πιστεύουν ότι δεν εννοούσαμε πολύ στα σοβαρά την νομοθεσία που υιοθετήσαμε, τότε έχουμε ε, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία, τη δημοσιονομική σταθερότητα και το μέλλον. Απειλή δεν είναι το να ακολουθούμε τους κανόνες, απειλή είναι το να γίνει δόγμα και πολιτική το να μην ακολουθούμε τους κανόνες. Και θα ήθελα να επισημάνω στην Κομισιόν ότι εσείς ε, υποχρέωση έχετε να φροντίσετε να ακολουθούμε τους κανόνες, όχι να του παραβιάζετε. Πολύ σύντομα, κυρία Κρέτσου. Ναι, θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι έχουμε έρθει εδώ για να δείξουμε ακριβώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενεργεί βάσει των κανόνων. Βεβαίως, δικαίως αναφέρεται ότι είναι η πρώτη φορά που ξεκινά αυτή τη διαδικασία. Όμως, θα ήθελα να σας πω ότι μπορείτε να βασίζεστε σε εμά και αύριο στο Σώμα των Επιτρόπων θα υπάρξει αυτή η ενημέρωση και δεν είναι προς το συμφέρον μας να κάνουμε περικοπές ή ε, να εφαρμόζουμε τυφλά τους κανόνες. Όμως, ταυτόχρονα, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο και πρέπει από κοινού να ενεργήσουμε ε, αν θέλουμε τα πράγματα να αλλάξουν. Σας ευχαριστώ γιατί μιλήσατε ακριβώς για αυτή την ε, κοινή επιμερισμένη ευθύνη μεταξύ ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Από κοινού λοιπόν θα πρέπει να ενεργούμε και όχι ε, να εκτοξεύουμε κατηγορίες για το τι είναι καλό μόνο στο εθνικό επίπεδο και το τι συμβαίνει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ Επίτροπη. Το πρώτο που θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε είναι ότι αυτοί που σε αυτό το κοινοβούλιο τοποθετήθηκαν κατά της αναστολής ε, των ε, κονδυλίων και φαίνεται ότι είναι ευρία πλειοψηφία, δεν ζητούν από την Κομισιόν να αγνοήσει ή να παραβιάσει τους κανόνες. Το μόνο που ζητούμε είναι η Κομισιόν να κάνει μια έξυπνη ερμηνεία των κανόνων που να εμποδίσει να ληφθεί μια άδικη απόφαση, αντιπαραγωγική απόφαση και που θα άφηνε την Κομισιόν σε μία θέση που θα ήταν ακατανόητη για τους πολίτες, δηλαδή να επιβληθεί τώρα μία κύρωση πιο σοβαρή από αυτό που έκανε σε σχέση με την ακύρωση των προστήμων. Κύριε Επίτροπη, είπατε ότι επιβάλλουν οι κανόνες την αναστολή των διαφορετικών ταμπίων. Όμως, κύριε Επίτροπη, υπάρχει κάποιος κανόνας που να θεσπίζει ένα ελάχιστο όριο της αναστολής των κονδυλίων και ουσιαστικά να εμποδίζει να είναι σε μηδενικό ποσό. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει αυτός ο κανόνας μεταξύ του μηδέν και του ανώτατου ορίου. Η Κομμασιόν έχει τη διακριτική ευθερία για να καθορίσει ένα ποσό και το τρόπο της αναστολής. Επομένως, κύριε Επιτροπή, αν έκανε μία πρόταση κομισιόν για την αναστολή των ταμείων, ε, να ήταν ένα ευρώ πάνω από το μηδέν δεν μπορεί να επικαλεστεί κανένα κανόνα γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κανόνας. Είναι μία απόφαση που λαμβάνεται από τη διακριτική ευχαίρεια της Κομισιόν και έρχεστε εδώ να μας πείτε ότι στην περίπτωση αυτή δεν έχετε περιθώριο λιγμών, ότι πρέπει να σεβαστείτε το κράτος δικαίου. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει ένας κανόνας που εμποδίζει τις μηδενικές κυρώσεις. Ξέρουμε όμως ότι δεν υπάρχει αυτό όταν η κυρία Μπέρες ρώτησε τους επιτρόπους αν θα μπορούσατε να σκεφτείτε μία μηδενική αναστολή και να προτείνετε αυτή τη λύση, ο κύριος Κατάινεν δεν είπε ότι αυτή η λύση θα ήταν ασυμβίβαστη με τους κανόνες, γιατί δεν είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες. Αυτό που είπε ήταν κάτι άλλο, ότι δεν ήθελε να προκρίνει την απόφαση της Κομισιόν, γιατί αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση η οποία μπορεί να λάβει η Κομισιόν στη διακριτική της ευχέρεια και μπορεί να εφαρμοστεί με έναν τρόπο έτσι ώστε να αποφευθεί μια άδικη απόφαση. κανόνες όπως έχουν υποχρεώνει στην Κομισιόν να ε, χρησιμοποιήσει τη διακριτική της ε, εξουσία και αρμοδιότητα έχοντας κατά νου την αρχή της αναλογικότητας και τον αντίκτυπο στις οικονομίες. Έτσι λοιπόν μην μας λέτε ότι δεν υπάρχει αντίκτυπος από την απόφαση αυτή, γιατί το επαναλάβατε πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτού του διαλόγου. Αναφερθήκατε σε ένα έγγραφο ε, το οποίο δημοσιεύτηκε στο πολίτικο και πράγματι εκεί έχει γραφτεί ότι η απόφαση δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στα, στις επενδύσεις και στα σημερινά έργα όμως ουσιαστικά έχει γραφτεί ότι μία απόφαση αναστολής θα καθυστερούσε τις επενδύσεις σαν να μπορούσαν οι οικονομίες αυτές δύο χωρών να μπορούσαν να υποστούν μια τέτοια καθυστέρηση και βασικά μόνο και μόνο η απειλή αυτή τη αναστολή ζημιώνει τι επενδύσει σε Ισπανία και Πορτογαλία. Είναι άδικη λοιπόν αυτή η απόφαση. κομισιών πρέπει εφαρμόζοντας τους κανόνες, δυνάμει των κανόνων να λάβει μια απόφαση δίκαιη για την Ισπανία και την Πορτογαλία και αυτή είναι η μη αναστολή των κονδυλίων. Κύριος Άλμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Μιλήσατε, κύριε Επίτροπε, για την εικόνα που θα δοθεί. Και επίσης ο Αντιπρόεδρος είπε ότι η Ισπανία μεγενθύνεται με εύρωστο τρόπο. Μια κομισιόν που έχει θετήσει την ανάπτυξη ως πολιτική στρατηγική, ποια αξιοπιστία θα έχει ή σε ποιο κίνδυνο μπαίνει να ζημιωθεί η αξιοπιστία της αν ε, ποινικοποιήσει την ανάπτυξη. Η Κομισιόν γνωρίζει τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό το θέμα στην εικόνα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, αν ε, τιμωρήσετε μία από τις χώρες, αν όχι τη χώρα που μεγεθύνεται περισσότερο στο σύνολο της Ευρωζώνης και τη χώρα που δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, τι εικόνα θα δώσουμε προς τα έξω τι μήνυμα θα δώσουμε στους πολίτες και από την άλλη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζα στο τελευταίο οικονομικό bulletin ουσιαστικά επενούσε τις προσπάθειες της Ισπανίας και της Γερμανίας στο εργοσιακό επίπεδο και παρότρινε και τις άλλες χώρες να ακολουθήσουν αυτήν την οδό. Ε, ποια αξιοπιστία θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν από τη μία επενεί τις μεταρρυθμίσεις μιας χώρας και από την άλλη την τιμωρεί τη χώρα αυτή η ερώτηση είναι γιατί μεγενθύνεται η Ισπανία, γιατί έκανα μεταρρυθμίσεις Βεβαίω, γιατί οι μεταρρυθμίσει που κάναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επιτυχεί επίση και λόγω τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, και λόγω των ενεργειακών τιμών. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριο λόγο είναι χωρί καμία αμφιβολία οι μεταρρυθμίσει, οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Και η ερώτησή μου είναι, αν είχαμε συμμορφωθεί αυστηρά με τους στόχους του ελλείμματος θα μπορούσαμε να έχουμε την εγγύηση ότι η Ισπανία θα γινόταν ακόμη περισσότερο από αυτό το 3,2% πιθανότατα όχι και πώς θα εξηγήσουμε στους πολίτες ότι θα τιμωρηθούμε ακριβώς γι' αυτό το λόγο και προσοχή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για να έχουμε μία βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη. Να μην ξεχνάμε ούτε αυτό το μέρος της συζήτησης που είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Ότι Αντιπρόεδρος Κατάινεν. Το έχω πει ξανά και ξανά, να τα ξαναπώ άλλη μία όμως. Βεβαίως δεν προδικάζουμε τα θα κάνουν και οι δύο χώρε αλλά και ε, η Επιτροπή. Ε, Ω συνομοθέτη, εσεί το Κοινοβούλιο, όταν υιοθετείτε νομοθεσία για εσά, δεν αποτελεί μια αφετηρία για δημιουργικέ ερμηνείε. Ο νομοθέτης επιθυμεί να συντάξει, να καταρτήσει ένα νόμο, ούτως ώστε όλοι να τον κατανοούν, να κατανοούν το πνεύμα αυτού του νόμου. Το πνεύμα του νόμου που θα πρέπει να γίνεται ευρέω, αποδεκτό και κατανοητό. Μόνο τότε έχει νόημα αυτό ο νόμο. Γι' αυτό και πολλοί, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες, πολλοί λοιπόν ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερμηνεύσει τους νόμους με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο τον κατέρτισαν αρχικά ε, οι νομοθέτες. Εμείς τον ερμηνεύουμε τον νόμο όπως έχει γραφτεί. Τους έχουμε ερμηνεύσει έξυπνα εντό εισαγωγικών, αλλά υπάρχουν και όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν κάτι δεν έχει αποκλειστεί, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εντάσσεται στο πνεύμα του νόμου. Και εδώ δεν μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο νόμο, αλλά γενικότερα. Εσείς λοιπόν ως νομοθέτες καταρτίζετε ένα νόμο και ε, με κάποιον τρόπο εμπεριέχεται και το πνεύμα του νόμου μέσα σε αυτή τη διατύπωση ανάμεσα στις γραμμές εντός εισαγωγικών. Μετά, για τον κύριο Σιλβιπερέρα. Θεωρείτε ότι οι δύο κυβερνήσεις θα υποβάλουν προσχέδιο προπολογισμού μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα συμμορφώνεται με τις ε, πιστώσεις, με τις δεσμεύσεις των ε, κυβερνήσεων. Εγώ το πιστεύω, γιατί είναι αναγκαιότητα. Είναι απαραίτητο για αυτές τις χώρες. Είναι απαραίτητο για την αξιοπιστία αυτών των χωρών, για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τις επενδύσεις. Υπάρχει λοιπόν ευρία στήριξη προς τις δύο κυβερνήσεις για να πράξουν το σωστό και απαραίτητο. Ιδάλλως ε, δεν ε, θα μπορέσουν να δρέψουν και τα ε, κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Σας ευχαριστώ. Μια πολύ σύντομη απάντηση, όχι τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Έκανε μια ερώτηση, Επίτροπος. Εγώ θέλω να επιβεβαιώσω, αλλά δεν είναι θέμα πίστης, δηλαδή να ξέρουμε αν η Ισπανία και η Πορτογαλία θα παρουσιάσουν τα σχέδια είναι πολιτικό το θέμα. Υπάρχει πολιτική δέσμευση από τις δύο κυβερνήσεις και δυστυχώς εδώ δεν... Συγγνώμη, ευτυχώς εμείς τώρα δεν ερχόμαστε να συζητήσουμε εδώ, αλλά ερχόμαστε να συζητήσουμε το περιεχόμενο της πρότασης που κάνει η Κομισιόν. Και αυτό το περιεχόμενο είτε είναι δίκαιο ή λογικό, είτε η Κομισιόν ε, ουσιαστικά παρουσιάζει κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε ε, στο επόμενο τμήμα της ε, συζήτησης. Τέσσερα λεπτά. Τέσσερα λεπτά. Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, Επιτροπή Προπολογισμού. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Προπολογισμών είναι κατά της αναστολής ε, των κονδυλίων των Διεθνικών και Επενδυτικών Ταμείων για την Πορτογαλία και την Ισπανία, η Κομισιόν και το Συμβούλιο ήδη αποφάσισαν να μην επιβάλλουν κυρώσει στην Πορτογαλία και την Ισπανία στα πλαίσια τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. Ήταν μια σωστή απόφαση που σεβάστηκε του ε, κανόνε, ε, την νομοθεσία, του κανονισμού και όλο το κοινοτικό κεκτημένο. Ήταν μια δίκαιη απόφαση απέναντι στι προσπάθειε που έκαναν οι δύο χώρε. Όμω όλοι γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια έγινε από τι τις οικογένειες, από τις επιχειρήσεις, από τους εργαζομένους, από τους νέους, από το πανεπιστήμιο, από τους αγρότες, ε, από τον ίδιο το λαό της Ισπανίας και την Πορτογαλίας. Μετά από την ορθή απόφαση να μην επιβληθούν κυρώσεις στα κράτη-μέλη, έχει κανένα νόημα τώρα να θέλετε να τιμωρήσετε τους πολίτες, τους δικαιούχους να, το να επιβάλλεται κυρώσεις στα κράτη, αυτό σημαίνει ένα πρόστιμο ενώ τώρα η αναστολή είναι πιο επιζήμια και τελικά πλήττει την οικονομία, την εμπιστοσύνη, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Εμεί ζητάμε σεβασμό των κανόνων, των αρχών, των κανονισμών και μόνο μία στάση μπορούμε να ακολουθήσουμε, να αποφασίσουμε για να μην εφαρμοστεί αυτή η αναστολή, γιατί θα ήταν άδικη και θα παραβίαζε την αρχή της ισότητας της μεταχείρισης των κρατών μελών. Ουσιαστικά είναι ε, υπάρχει κάτι παράλογο. Αν η Πορτογαλία ε, είχε σεβαστεί το πρόγραμμα θα βρισκόταν σήμερα στο δεύτερο πακέτο διάσωσης εδώ. Αυτό που μπορούμε ε, να κάνουμε είναι το εξής. Θα πρέπει να δούμε πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες. Η Κομισιόν μέσω της προσαρμογής ξέρετε πολύ καλά κύριε Επίτροπε τι έγινε με την τεχνική προσαρμογή και για τις άλλες χώρες ε, με την Ιταλία, με την Ισπανία ε, είχαμε ε, ουσιαστικά για πάνω από ένα δισεκατομμύριο αναλήψεις υποχρεώσεων και μιλάτε τώρα για την Ισπανία αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων δεν έχει νόημα αυτό έτσι λοιπόν εσείς αναφέρατε ότι η αναστολή δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην εκτέλεση των προγραμμάτων. Αυτό είναι ψευδές. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι δύο επίτροποι ξέρουν τη διαφορά μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών. Για να έχουμε πληρωμές, καταρχήν πρέπει να έχουμε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Οι πληρωμές είναι συνέπεια των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων. Αν παγώσετε και να στείλετε όλες τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, δεν θα λάβει χώρα καμία πληρωμή. Και εμεί μιλάμε για νέα σχέδια, για νέα έργα. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας ε, και ξέρετε είναι ε, ουσιαστικά πρωταθλητής στην εκτέλεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων η Πορτογαλία. Δεν είχε πολύ μεγάλο κονδύλι και αν ε, δείτε την ικανότητα απορρόφησης το 2016 έχει τρία εκατομμύρια πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Αυτά τα χρειάζεται η πορτογαλική οικονομία. Εγώ ξέρω ότι η Επίτροπος θέλει εξαιρετική εκτέλεση των πιστώσεων, όμως ε, είναι ε, χείριστη η εκτέλεση των κονδύλιων της πολιτικής συνοχής. Κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να ξέρετε ότι η αναστολή των ανλήψεων υποχρεώσεων προκαλεί πρόβλημα στις πληρωμές τα επόμενα χρόνια. Δεν θα υπάρχουν πληρωμές. Έτσι λοιπόν, εγώ αυτό που περιμένω είναι η Κομισιόν να αποφασίσει να μην αναστείλει ε, τα κονδύλια. Γιατί το αντίθετο θα ήταν ένα τεράστιο πολιτικό λάθος και για μας θα έχριζε της μεγίστης λογοκρισίας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ακούσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι σαφέστατα όλα όσα υπόθηκαν εδώ. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος θα σας δώσω το λόγο. Εντάξει, θα επιδείξω ευελιξία. Ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το ίδιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Απλά ήθελα να πω ότι σα είδα ήδη από την αρχή ότι το μέτρο αυτό δεν έχει, κανέ, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που έχουν χειριστεί οι χώρες αυτές ε, τα ταμεία. Και θα θυμάστε ότι η πρώτη μου ε, ε, επίσκεψη ήταν στην Πορτογαλία. Θέλω να τη συγχαρώ επειδή ήταν η πρώτη χώρα που απορρόφησε όλα τα χρήματα από το πρόγραμμα ε, για το 2017 έως 2013. Ε, δεν έχει καμία σχέση με το πώς ε, λειτουργούν τα πράγματα επιτόπου. Και όπως σας είπα, η Πορτογαλία είναι πολύ καλός μαθητής, όπως είπατε. Thank you for Committee Ευχαριστώ πολύ. Η Σοφία Ριπέιρο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εμείς ε, από την Επιτροπή Επασχόλησης θέλουμε να πούμε ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι σε οποιαδήποτε αναστολική περικοπή των ταμείων για την Πορτογαλία και την ε, Ισπανία. Αυτό εκφράζεται και στο έγγραφο που εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι εντελώ και σοφρονική κατάσταση που ζούμε. Αυτέ ε, οι χώρε δεν έχουν σεβαστεί, κάποιε χώρε δεν έχουν σεβαστεί κάποιε από τι δεσμεύσει. Όμω ακόμη δεν έχει τελειώσει η προθεσμία ε, για τις χώρες αυτές. Ο Επίτροπος Κατάινεν και το 2015 είπε η Πορτογαλία έκανε ένα θαύμα τρία χρόνια αφού μπήκε στο πρόγραμμα, επέστρεψε στην ανάπτυξη και σταθεροποίησε την κατάσταση. Όμως οι περικοπές της επενδύσεις δεν είναι συμβατές με την ανάπτυξη και υπάρχει... Ε, δεν υπάρχει τρόπος για ήπια εφαρμογή, όμως ε, υπάρχουν ε, ε, κάποια κονδύλια πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλα τα κονδύλια προωθούν την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, είτε μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις εργασίες και να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Δεν μπορούμε να στερήσουμε ε, από τις χώρες αυτές την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όταν τη χρειάζονται περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή κάνει σαν ένα γιατρό που εξηγεί στον ασθενή του να πάρει τα φάρμακα και τα ωφέλη αυτών όμως κατόπιν δεν συνταγογραφεί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε είμαστε πολιτικοί ή τεχνοκράτε Αν συνεχίζουμε να ε, εφαρμόζουμε τεχνοκρατικά μέτρα ή αν ε, θα ε, φροντίσουμε έτσι ώστε αυτά τα μέτρα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Εδώ θα έχουμε δύο συνέπειες ή θα συνεχίσουμε να μεγενθύνουμε το χάσμα μεταξύ των πολιτών και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ή θα προωθήσουμε αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτή η απόφαση δεν θα θίξει και θα πλήξει μόνο την Πορτογαλία και την Ισπανία αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριο Σέρτζιο κύριε Πρέτο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και ο Επίτροπο στη θέληση του Ευρωπαίου Νομοθέτη. Εγώ ήμουν ε, από τους Σοσιαλιστέ στην αναθεώρηση του κανονισμού ε, για τα ε, ταμεία πριν κάποια χρόνια και ήμασταν πάρα πολύ επικριτικοί όταν ε, εισήχθη η μακροοικονομική ρεσιμότητα και θέλαμε μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Γιατί, γιατί πιστεύουμε ότι ήταν απαραίτητο στην πολιτική συνοχής, ε, η πολιτική συνοχής να υπερισχύει της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ε, η ε, πολιτική συνοχής δεν είναι ένα εργαλείο ε, για την μακροοικονομική διόρθωση. Εμείς τώρα εδώ μιλάμε για το πώς θα πρέπει να γίνει η ερμηνεία των κανόνων και εγώ σας λέω ως νομοθέτης ότι υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών για να είναι μηδενικές οι κυρώσεις. Τώρα, αν εμείς ε, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, ε, εσείς όμως μας λέτε ποιος είναι ο πολιτικός στόχος που επιζητούμε τη στιγμή της αναστολής των κονδυλίων. Γιατί αν ο πολιτικός στόχος είναι το να ε, πληρωθεί ο στόχος του ελλείμματος, ε, τότε ουσιαστικά το να αναστείλουμε τα κονδύλια θα απομακρύνουμε τις χώρες από την επίτευξη του στόχου αυτού, γιατί θα πλήξουμε πάρα πολλές μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Αν ο πολιτικός στόχος είναι, εσείς ε, φαίνεται να τραβήξετε το αυτές τις κυβερνήσεις για να συμμορφωθούν με τον πολιτικό στόχο, εγώ σας είπα να είστε σκληροί στις δηλώσεις τους, αλλά να μην είστε σκληροί με τους πολίτες που θα έρθουν να πληρώσουν το λογαριασμό. Γι' αυτό εγώ λέω ότι υπάρχει περιθωρίο λιγμών αν υπάρχει πολιτική βούληση. Εσείς ε, μπορείτε να σεβαστείτε το άρθρο 12γ που λέει όταν η επιστροφή βλέπει ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα για τη διόρθωση του ελλείμματος μπορούν να ανασταλούν οι κυρώσεις. Στην περίπτωση της Ισπανίας με την πρόταση που έκανε περίπτωση χάρη η Ισπανική κυβέρνηση για τον εταιρικό φόρο. Δεν χρειάζεται εσείς ε, στις 15 Οκτωβρίου ε, να αναλάβετε δράση. Αν έχετε πολιτική βούληση ήδη το άρθρο 23 σας δίνει την ευελιξία για να είστε όχι μόνο ευέλικτη αλλά και δίκαιη με τους πολίτες και φυείς. Ευχαριστώ για την Επιτροπή Άγκρη. Αγγιέρα Γκαρσία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Κατάινεν σε μια ερώτηση που έκανε πριν. Ο νόμος είναι για να τον σεβόμαστε φυσικά ε, όλοι οι νόμοι και οι υποχρεώσει είναι για να τι σεβόμαστε. Το ίδιο ισχύει και με την ερασιμότητα. Όμως, Επίτροπε Κρέτσου, δεν ε, μπορούμε ε, τουλάχιστον από τα αριστερά εμείς οι σοσιαλιστές να θεωρούμε ότι είναι αυτό ένας κανός που μας κάνει περήφανος. Πρέπει όμως να το σεβαστούμε και στη συνέχεια εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι ίδιο σε όλες οι καταστάσεις. Ακόμα και αν σεβαστούμε τους κανόνες είναι άνισες οι καταστάσεις εδώ ε, μιλάμε για μια κυβέρνηση ε, που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της και είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση η χώρα μου και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Ε, δηλαδή έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε και τι συμβαίνει με την ανεργία. Θέλω να μιλήσω και τι συμβαίνει με το Ταμείο της ε, αγροτικής ανάπτυξης. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στην Ισπανία, τα 17 προγράμματα δεν έχουν εγκριθεί παρά ε, λιγότερο εδώ και λιγότερο από ένα χρόνο και ακόμη δεν έχουν μπορέσει να δεθούν σε εφαρμογή αυτά τα προγράμματα και από ό,τι φαίνεται ότι το πρόγραμμα ΦΕΝ εγκρίθηκε λιγότερο από 9 μήνες πριν και δεν έχει φτάσει ακόμα στις περιφέρειες. Έτσι λοιπόν ε, ουσιαστικά Έχουμε δύο ταμεία πάρα πολύ σημαντικά για την ε, ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν η απόφασή σας ε, σχετίζεται πάρα πολύ με αυτά. Ε, κοιτάξτε, Έχουμε τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής και εκεί αποφασίστηκε ένα μηδενικό ποσοστό και δεν άλλαξε για τρία χρόνια αυτό το ποσοστό λόγω μιας έκτασης εξαιρετικής κατάστασης. Σκεφτείτε λοιπόν εσείς τις αναγκαιότητες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, σεβόμενοι τους κανόνες. Αυτό σας ζητώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ζωνομέλο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπη προφανώς αναστολή ε, είναι τιμωρία και δεν το αξίζει η Πορτογαλία. Μία χώρα η οποία μείωσε το έλλειμμά της που ήταν 11% ε, το 2010 και 3% το 2015, το εν αξίζει να τιμωρηθεί, αλλά αξίζει επένους. Εγώ αυτό έχω κατά νου. Εσείς ουσιαστικά τιμωρείτε τον καλό το μαθητή. Και αυτό τι σημαίνει τελικά ότι κάποιος κάνει προσπάθειες και δεν ανταμείβεται. Εγώ ήθελα να ζητήσω η Επίτροποι να μην δώσουν λιγότερα στην Περτογαλία πόσο ο Επίτροπος ε, Πιέρ Μοσκοβισή και ο Γάλλος Υπουργών ε, οικονομικών αποφάσεων για την Γαλλία και έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013. Ο κ. Μοσκοβισή ε, είχε υποσχεθεί έλλειμμα 3% ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτευχθεί ο στόχος και ο Επιτροπός ε, ε, ε Πιέρ Μοσκοβισή ζήτησε ε, περισσότερο χρόνο. Ξέρετε ποιο είναι τώρα το 2015 η πρόβλεψη του κυρίου Μοσκοβισή για τη Γαλλία 2%. Ενώ ξέρετε τι συνέβη στα τέλη του 2015 στη Γαλλία 3,2%. Ε, και ο Υπουργός Οικονομικών δεν είναι εδώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στην Πορτογαλία και στην Ισπανία δεν έχουν να κάνουν ε, ε, ουσιαστικά με το τι εφαρμόστηκε στη Γαλλία. Δηλαδή δεν μπορείτε να τιμωρείτε την Πορτογαλία ε, και την Ισπανία για τους ίδιους λόγους που δεν τιμωρήσατε τη Γαλλία. Εγώ ξέρω ότι δεν επιβάλλατε κυρώσεις στη Γαλλία γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ανταμείβει τις προσπάθειες εμείς ε, έχουμε ζητήσει πάρα πολλές θυσίες από τους εργαζομένους, από τους λαούς, ε, από τις οικογένειες. Η Πορτογαλία εφάρμοσε το πρόγραμμα διορθωτικών προσαρμογής, διορθωτικής προσαρμογής ε, μέσα σε ένα χρονικό όριο που είχε προβλεφθεί από την Κομισιόν. Και δεν ήταν κάτι έκτακτο που καμία ε, ουσιαστικά κυβέρνηση, αν δεν ήταν μάλλον μια έκτακτη περίπτωση όπως έγινε στην περίπτωση της Μπανίφ που δεν μπορούσε να το προβλέψει η κυβέρνηση, δεν θα είμαστε τώρα ε, σε αυτή την κατάσταση. Εσείς ε, για τη Γερμανία ουσιαστικά απαιτήσατε τα ίδια πράγματα που μιλάτε σήμερα από την Πορτογαλία και την Ισπανία για να μην μιλήσω και το τι έγινε με τη Φιλανδία. Ευχαριστώ. Και τέλος, πρωτού δώσουμε τον ε, λόγο στους επιτρόπους, Αλέν Καντέκ, πρόεδρος της Επιτροπής ΠΕΣ, για τέσσερα Ευχαριστώ. Ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Αλληλείας μιλώ εδώ, αλλά και ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας. Είναι ένα ταμείο το οποίο αφορά άμεσα την Πορτογαλία και την Ισπανία και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό το στοιχείο. Επίση πρέπει να πω ότι είμαι αντίθετο, κάθετα αντίθετο στην αναστολή των ε, ταμείων, γιατί εδώ πρόκειται για ένα ε, μέτρο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά για τι δύο αυτέ χώρε. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τι κοινωνικο-οικονομικές ε, περιστάσεις και συνθήκε σε κάθε χώρα. Αυτό αναφέρεται στον κανονισμό. Εγώ πρέπει να πω ότι αισθάνομαι και Πορτογάλος και Ισπανός. Και δεν είναι η στιγμή, η κατάλληλη ώρα να ε, κάνουμε τέτοιες ε, επιλογές. Πολιτικά θα είναι καταστροφικό και για την Ισπανία, για την Πορτογαλία, αλλά και για την Ευρώπη ευρύτερα. Ήδη οι πολίτε έχουν απομακρυνθεί από την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να ενισχύσουμε αυτή την απομάκρυνση. Ε, και επενείται την Πορτογαλία, αλλά και προτείνεται να την τιμωρήσετε, κυρία Επίτροπε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι ακριβώ συμβαίνει. Είμαι κάθετα αντίθετο σε αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτή η Επιτροπή τυφλά ε, τηρεί τους κανόνες χωρίς καμία ερμηνεία. Μάλιστα, για το αντίθετο μας έχουν κατηγορήσει. η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν έλαβαν πρόστιμο ακριβώς επειδή εξοποιήσαμε αυτό το περιθώριο ελιγμών ε, με την ε, έξυπνη ερμηνεία των νόμων. Λάβαμε υπόψη και την πολιτική κατάσταση και την οικονομική κατάσταση. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία τυφλή εφαρμογή των κανόνων θεωρούμε ότι οι δύο κυβερνήσει ε, ε, κάνουν ό,τι μπορούν ε, κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε. Και είμαι βέβαιο ότι και εσεί είστε πλήρω ενήμεροι σε ό,τι αφορά το μέγεθο των αναξιοποίητων πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμών. Ανεξάρτητα από την απόφασή μας για το θέμα της αναστολής. Υπάρχει όμως ε, κοινή, επιμερισμένη ευθύνη. Πρέπει λοιπόν και τα κρατημέλη να ε, αναλάβει το καθήκον της και η Ευρωπαϊκή Ελληνική το δικό της. Κάποιες ε, παρεμβάσεις ανέφεραν το... Μάλλον παρουσίασαν μια σύγχυση σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την αιρεσιμότητα. Θα σταματήσω λέγοντας μόνο κάτι τελευταίο, μια προσωπική νότα. Ήμουν υπουργό ε, Οικονομικών όταν ε, είχαν εγκριθεί όλα τα πακέτα ε, δημοσιονομικής ενίσχυσης και διάσωση. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο γιατί τα κράτη-μέλη δεν εμπιστεύονταν το ένα το άλλο. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε καμία συμφωνία για το πώς θα βοηθήσουμε τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εν μέσω κρίσης δημιουργήσαμε ένα σύστημα το οποίο θεωρήθηκε δίκαιο από όλους. Τώρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο δίνει ένα νομικό πλαίσιο ε, προς την Επιτροπή για να εφαρμόζει ε, τους ίδιους κανόνες σε όλα τα κρατημέλη. Είμαι βέβαιος ότι η μία κέρια, θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αλληλεγγύη. Όμω, και ο κόσμος θα πρέπει να έχει την εντύπωση ότι και το πολιτικό μας, το συνομινομικό μας σύστημα είναι δίκαιο. Γι' αυτό όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερμηνεύει τους κανόνες πρέπει να μεριμνεί ώστε να μην βρίσκουμε μόνο τρόπους να παρακάμψουμε το πνεύμα του νόμου, αλλά να τηρούμε τους κανόνες με σωστό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, συνθήκες, αλλά να τηρούμε και τους κανόνες που είναι βιώσιμοι και μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Ε, για μένα ήταν πολύ θετική εμπειρία. Όπως ξέρετε έχουμε στείλει και επιστολή στο Κοινοβούλιο πριν από δυόμιση μήνες και είμαστε πάντα διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ, η Επίτροπος Κρέτσου. Θα ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω και εγώ για αυτή την ε, πολύ ανοιχτή συζήτηση, πολύ ειλικρινή, για ένα πολύ δύσκολο και καθόδε ζήτημα είναι όντω ε, δύσκολο, όμω ε, πρέπει ταυτόχρονα να πούμε ότι αυτοί είναι οι κανόνες. Για το τελευταίο ερώτημα που έλαβα, δεν είναι αν εγώ ή ο αντιπρόεδρος Κατάνια να αποφασίσαμε κάτι, απλώς ακολουθούμε του κανόνες. Όταν ο κύριος Βανίσταν ρωτή είπε στην αρχή ήδη ότι ήταν μια ε, δύσκολη συζήτηση και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου το θέμα της αιρεσιμότητας. Κάποια μέλη το υπερψήφισαν και είπαν ότι πρόκειται για θετική αιρεσιμότητα. Ας δούμε λοιπόν από κοινού πώς μπορούμε ε, να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία και όχι για να κατηγορούμε ότι είμαστε πολύ καλοί για κάποια κράτη-μέλη και ε, πολύ αυστηροί με άλλα. Ε, αύριο ε, στο Σώμα των Επιτρόπων θα μεταφέρουμε τις απόψεις σας και βεβαίως το Σώμα θα αποφασίσει. Είμαι βέβαιη όμως ότι και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ε, και της διάσκεψης των Προέδρων θα μάλλον των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, θα δημοσιεύσει μία ανακοίνωση. Να είστε βέβαιοι ότι αύριο εγώ θα μεταφέρω τα όσα μου είπατε στους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω και εγώ ότι ήταν πολύ ε, χρήσιμος ε, και ζωντανός ο διάλογος και σημαντικός. Όπως είπαμε στην αρχή της συνεδρίασης αυτής, η σημερινή συνάντηση δεν κλείνει απαραίτητα τον διάλογο αυτό και θα πρέπει καταρχάς να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι καμία απόφαση δεν μπορεί να υιοθετηθεί επίσημα πριν από την ολοκλήρωση του διαφρομένου διαλόγου. Οι συντονιστές στο Προεδρείο θα αποφασίσουν ε, θα, θα υποβάλουν σύσταση στην διάσκεψη των Προέδρων η οποία θα αποφασίσει εάν δηλαδή θα υπάρξει συγκεκριμένη γνωμοδότηση ή εάν το Κοινοβούλιο ζητήσει να παρατείνει τον διαρθωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι αυτό ακολουθεί και το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Πρώτη διευκρίνηση ήταν αυτή. Η δεύτερη είναι ότι διαπιστώσαμε ότι μπορεί να έχουμε διαφορετική ερμηνεία όσον αφορά το πνεύμα του νόμου. Νομίζω όμως ότι η συζήτηση αυτή αποτελεί ένα βήμα προοδού, διότι το γράμμα του νόμου μπορεί να αποτελεί υποχρέωση ε, ε, ε, ανάληψης δράσης, δεν προβλέπει όμως κάποια συγκεκριμένη προθεσμία. Μπορεί να διαφωνούμε λοιπόν όσον αφορά το πνεύμα του νόμου. Αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν και τελευταία παρατήρηση. Εγώ θα περίμενα και δεν θέλω να κατηγορήσω την Κομισιόν, αλλά περίμενα πιο συγκεκριμένα να μου πει τι πρόταση θα υπέβαλε, δηλαδή τι ποσό για ποιο πρόγραμμα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε το διάλογό μας. διότι δεν έχω δει ακόμα συγκεκριμένα ονόματα προγραμμάτων ε, και αριθμητικά στοιχεία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δίνω το λόγο στη Συμπρόεδρο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα λόγια. Επιτρέψτε μου. Διαδικαστικό. Διότι δεν θα συμμετάσχω στην ε, συνεδρία των συντονιστών. Στα πορτογαλικά, επιτρέψτε μου. Ε, Εγώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, έκανα ένα αίτημα και στις δύο επιτροπές ε, βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού 2011 στο ότι η κυβέρνηση της ε, Πορτογαλίας να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη διάταξη του κοινωνισμού ότι οι επιτροπές μπορούν, είναι μια διευκόλυνση, να καλέσουν τα κράτη προορισμού των μέτρων να συμμετέχουν στον διαθροτικό διάλογο. Εγώ είμαι νομικός και ξέρω ε, ουσιαστικά τα πράγματα αυτά και θα ήθελα να πει η χώρα μου ε, ουσιαστικά αυτό που θεωρεί ότι είναι σωστό. Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι κι άλλοι θα θέσουν αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ναι, είναι σαφές για όλους εμάς αυτό, σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, όλα τα μέλη και των δύο επιτροπών για τον ειλικρινή διάλογο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επειδή κατανοείτε την ευθύνη μας να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες κάθε μία από τις πράξεις μας εδώ στο Κοινοβούλιο και από κοινού και με την Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τα επόμενα βήματα, θα ήθελα να καλέσω τους συντονιστές των δύο επιτροπών και τα Προεδρία των δύο επιτροπών να παραμείνουν σε αυτή την αίθουσα και κλεισμένων των θυρών και να αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε με τον δευρωμένο διάλογο, γιατί όλοι μας κατανοούμε ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα του διαλόγου. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, και συνεχίζουμε. Ολοκληρώνω τη συνεδρίαση.